κύριοι. Θα συνεχίσω στα πολωνικά, λέει ο πρόεδρος. It's okay with translation? Yes, yes. It's okay. Porządek dzisiejszego posiedzenia został... Έχετε μπροστά σας το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Έχετε παρατηρήσεις παρακαλώ. Όχι από ό,τι βλέπω. Οπότε θα ήθελα τώρα να υπογραμμίσω ότι δεδομένου ότι η πρόεδρός μας συμμετέχει σε μια αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη στον ΟΗΕ, σήμερα θα πρέπει να ικανοποιηθείτε με τη δικιά μου Προεδρία. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε καρποφόρα κατά τη διάρκεια ολόκληρης της σημερινής ημέρας. Έχετε λοιπόν το σχέδιο ημερήσιας διάταξης μπροστά σας. Έχουμε την ώρα των ερωτήσεων, μετά θα ασχοληθούμε με την Νοτιοανατολική Ασία, Ινδονησία πιο συγκεκριμένα, μετά θα ασχοληθούμε με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βερμανία. και σήμερα το απόγευμα θα έχουμε εδώ τον κύριο Ποπόφσκι. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με την Αίγυπτο. Στις 4.30 ε, θα μιλήσουμε για τη Ζουαζιλάνδη και μετά για την ε, Βόρεια Κορέα και στη συνέχεια για την Κινέα Κόνακρη. Έχουμε λοιπόν πολλά θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε σήμερα. Ελπίζω να μπορέσουμε να τα εξετάσουμε όλα σε βάθος. Το δεύτερο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έγκριση των πρακτικών τη συνεδριάσεώ μα τη 3η και 4η Οκτωβρίου 2011. Έχετε σχόλια, παρατηρήσει. Όχι. Συνεπώ θεωρώ ότι εγκρίνονται τα πρακτικά αυτά. Έρχομαι τώρα στι ανακοινώσει του Πρόεδρου. Θέλω να σα υπενθυμίσω ότι στην προηγούμενη, στην τελευταία μας ολομέλεια εγκρίναμε ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρώτα απ' όλα για το Ιράν πρόκειται για την μη τήρηση των μη σεβασμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Διαπιστώνουμε ότι γίνονται όλο και περισσότερες συλλήψεις ακτιβιστών υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι παρατηρείται επίσης ε, ε, πρόβλημα με τη δικαιοσύνη, ότι διώκονται οι μειονότητες, διώκονται όσοι μάχονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι δικηγόροι, οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Δυστυχώς έχουμε και πάρα πολλές περιπτώσεις εκτελέσεων στο Ιράν. Η θανατική ποινή ε, δυστυχώς ε, αποφασίζεται και ε, σε περιπτώσεις ανηλίκων. Δεν υπάρχει μορατόριο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει ένα μορατόριο για να μην υπάρχουν άλλες θανατικές ποινές. Στη συνεπόμενη συνεδρίασή μας, στις 5 Δεκεμβρίου δηλαδή, θα μιλήσουμε με έναν ειδικό εκπρόσωπο του ΟΗΕ, τον κύριο Σακή, ειδικό για το, για το Ιράν. Και ελπίζω να μπορέσουμε να βαθύνουμε περισσότερο σε αυτό το θέμα. Επίσης είχαμε και ένα άλλο ψήφισμα για τον κύριο Αλά Αμπτελ Φατά, που είναι ο blogger στην Αίγυπτο. Ε, ζητάμε να απελευθερωθεί αμέσως ε, και να βγει από τη φυλακή ο blogger αυτός. Ζητάμε από τις αρχές της Αιγύπτου να μην φέρνουν σε στρατιωτικά δικαστήρια ε, πολίτες Δυστυχώ είναι μια πρακτική που ακολουθείται πολύ συχνά στην Αίγυπτο. Θα το συζητήσουμε αυτό σήμερα όταν φτάσουμε στο σημείο εκείνο όπου θα εξετάσουμε τη σημερινή κατάσταση στην Αίγυπτο. Φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας αυτή. Τώρα, στις 28 Νοεμβρίου στην ε, Ουάσιγκτον υπάρχει η διάσκεψη κορυφής Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ένα ψήφισμα για το θέμα αυτό, με το οποίο κάνει έκκληση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των δύο αυτών ε, υπήρων με στόχο την ειρήνη. Μιλάμε επίσης για το εμπόριο, για τις επενδύσεις, για την αύξηση θέσεων απασχόλησης και ζητήσαμε επίσης να επαναληφθεί ο διάλογος ανάμεσα στους Παλαιστινίους και το Ισραήλ. Στηρίζουμε την επιθυμία των Παλαιστινίων να εκπροσωπούνται στον ΟΗΕ, είναι, να έχουν αντιπροσωπεία δηλαδή στον ΟΗΕ, γιατί είναι κάτι ε, το οποίο ενθαρρύνει τις δημοκρατίες που σιγά σιγά εμφανίζονται στην Αφρική, τις ενθαρρύνει να συνεχίσουν. Επικρίνουμε επίσης το Ιράν και τον κίνδυνο που αποτελεί η χώρα αυτή που θέλει να έχει πυρηνικά όπλα. Ε, έχουμε επίσης και ένα ψήφισμα για την Ουκρανία. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 17 Νοεμβρίου ενέκρινε ένα κείμενο όσον αφορά τις Συμφωνία σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας. Εμείς θέλουμε οι διαπραγματευτές από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουν ό,τι προσπάθειες μπορούν προκειμένου η συμφωνία αυτή να ολοκληρωθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα. Το καλύτερο θα ήταν η υπογραφή αυτή να λάβει χώρα φέτος ακόμα. Αλλά όπως έχουμε επίσης υπογραμμίσει, θα πρέπει όλα αυτά ε, να γίνουν σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου. Στο ψήφισμα αυτό εμείς σημειώνουμε ότι η το ότι δεν καταδικάζεται το γεγονός ότι βρίσκεται η Γιούλια Τιμωσέγκο στην φυλακή μπορεί να αποτελέσει ένα εμπόδιο. Επίσης ενημερωθήκαμε για την κατάσταση υγείας της Γιούλια Τιμοσέγκο και μάθαμε ότι υπάρχουν προβλήματα και έχουμε λάβει πάρα πολλά αιτήματα που ζητούν την απελευθέρωση της κυρίας Τιμοσέγκο. Το 25 Νοεμβρίου γιορτάσαμε την ε, Διεθνή ημέρα για την καταπολέμηση της ε, βίας βάρος των γυναικών. Ανταλλάξαμε απόψεις με διάφορους εκπροσώπους, για παράδειγμα από το Κονγκό, την Λιβερία και το Αφγανιστάν. Οι γυναίκες από τις χώρες αυτές μας παρουσίασαν τις δικές τους εμπειρίες, τι πέρασαν δηλαδή κατά τη διάρκεια ένοπλων σειράξεων στις χώρες τους. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θεωρεί τις ε, ε, βιότητες, τις σεξουαλικές αυτές, μια πρακτική πολέμου που επίτηδες ε, λαμβάνει χώρα ως τακτική πολέμου. Για πρώτη φορά λοιπόν μπορούμε να καταδικάσουμε αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν την τακτική αυτή. Εγκρίναμε επίσης κείμενο το οποίο καταδικάζει την ενδοοικογενειακή βία. Αυτό αποτελεί τεράστια πρόοδο σε σχέση με την κατάσταση όπως είχε πριν από 10 χρόνια. Βέβαια εννοείται ότι μας μένει ακόμα αρκετός δρόμος. Φαντάζομαι ότι αυτό το θέμα θα το θίξουμε ξανά και ξανά στο μέλλον. Επίσης, έχουμε πολλά ζητήματα να λύσουμε σχετικά με την βία αυτή σε βάρος των γυναικών. Μιλήσαμε μιλήσ, επίσης για τον Άλεξ Γκαλάσκι, που είναι ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ήρθε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μίλησε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων τον Ιούνιο που μας πέρασε. Και ακριβώς, αλλά εδώ μιλάω εκ μέρους του αυτού μου και μόνο, πιστεύω ότι η ομιλία του αυτή είχαν σαν αποτέλεσμα οι αρχές της Λευκορουσίας να αναλάβουν ε, δράσεις πολύ αυστηρές σε βάρος του. 24 Νοεμβρίου, για παράδειγμα, καταδικάστηκε σε 4,5 χρόνια ε, καταναγκαστικά έργα. Τον ε, κατηγόρησαν ότι έκρυβε τα έσοδά του, τα οποία ήταν παράνομα και σε αυτό βασίζεται η καταδίκη του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσίευσε μια ειδική δήλωση από αυτού στον τύπο. Αυτό όσον αφορά τα πιο πρόσφατα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πιο συγκεκριμένα της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε στο σημείο 4. Πρόκειται για τις ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση είναι της κυρίας Νίκολσον. Νικόλ Κιλ Νίλσερ, μάλλον. Και μετά η κυρία Μπρισπέρο. Φρίντα Μπρίπουλς. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα με την πρώτη ερώτηση. Της κυρίας Κιλ Νίλσεν, για την οποία θα μιλήσει η κυρία Μπρέπουλς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η Νικόλ, η συνάδελφός μου, μου ζήτησε να αναλάβω εγώ την ερώτηση αυτή. Δεν είναι ότι βρίσκεται στην Νέα Υόρκη, απλώς θα έρθει αργότερα από τη Γαλλία δεν μπορεί να είναι εδώ ακόμα. Είναι ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται... Πρόκειται για μια ειδική μορφή βασανισμού σε βάρος γυναικών. Η ερώτηση είναι... Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα βασανιστήρια. Με ποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν μπορεί να μας διαβεβαιώσει ότι η διάσταση του φύλου στους βασανισμούς θα λαμβάνεται ικανοποιητικά υπόψη στις κατευθυντήρες αυτές γραμμές δηλαδή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Μισελσούν θα απαντήσει στην ερώτηση αυτή από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε παραδείγματα βασανισμών, όπως αυτά που αναφέρονται στην ερώτηση της κυρίας Νίλσεν βιασμοί, βασανιστήρια σε βάρος γυναικών κλπ. Ουσιαστικά τα εξετάζουμε αυτά στα πλαίσια άλλων κατευθυντηρίων γραμμών, που είναι η βία ε, σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών. Το Συμβούλιο δουλεύει πάνω σε αυτό το θέμα και ενέκρινε πρόσφατα μία σειρά περιφερειακών προτεραιοτήτων στα πλαίσια των κατευθυντηρίων αυτών γραμμών που περιλαμβάνουν την περίπτωση των καταναγκαστικών ε, γάμων, των γάμων που γίνονται με πολύ νέα κορίτσια. Ε, πρόκειται για την ε, συμμετοχή στα πολιτικά των γυναικών. Πρόκειται επίσης για τους ακροτηριασμούς σε βάρος γυναικών. Πρόκειται για τους βιασμούς σε περιπτώσεις πολεμικών σειράξεων, είναι αυτά πράγματα τα οποία βρίσκονται στο πρόγραμμά μας για του χρόνου. Συνεπώς, όσον αφορά την ουσία, το εξετάζουμε το θέμα αυτό κάτω από διαφορετικούς τίτλους, σε πολλά σημεία δηλαδή της πολιτικής μας, αλλά όπως και να έχει το πράγμα, υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές για τα βασανιστήρια και Ολοκληρώνεται η διαδικασία αυτή την εποχή σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κοινωνία των πολιτών. Ο στόχος μας είναι πάντα να μπορούμε να επηρεάζουμε τις τρίτες χώρες να παίρνουν αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση των βασανισμών. Γι' αυτό και υπάρχει ένα ειδικό κεφάλαιο στις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρεται σε ομάδες που απαιτούν ειδική προστασία. Εκεί ενθαρρύνονται τρίτες χώρες προκειμένου να αποφασίσουν για προδιαγραφές τέτοιες οι οποίες θα προστατεύουν μεταξύ άλλων και τις γυναίκες οι οποίες ε, απαιτούν ειδική προστασία από βασανισμούς και διότητες. Όπως σας είπα, μετά την διαβούλευση καταλήγουμε αυτή την εποχή και έτσι αυτά είναι τα δύο πακέτα κατευθυρίων γραμμών που έχουμε για το θέμα της προστασίας των γυναικών από τα βασανιστήρια. Ελπίζω έτσι να έχω απαντήσει στην ερώτηση. Ευχαριστούμε. Κυρία Μπρίπουλς, έχετε κάτι να προσθέσετε. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις πληροφορίες που μας δίνει. Είναι όντως πολύ σημαντικό και για τη συνάδελφο και για όλους μας. Η προβληματική δηλαδή να παραμένει, είτε πρόκειται για αυτές τις κατευθύνες γραμμές, είτε για άλλες, να υπάρχει αυτή η προβληματική που μας απασχολεί. Το σημαντικό είναι τα δύο πακέτα κάποια στιγμή να συγχωνευθούν και κάποια στιγμή να καταλήξουν στον ίδιο στόχο. Είναι μια σαφής απάντηση. Εμείς θα παρακολουθούμε τι θα γίνει από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσο μπορούμε περισσότερο, θα παρακολουθούμε τη συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα περνάμε στην επόμενη ερώτηση που είναι η νομοθεσία του Ισραήλ σχετικά με τη λειτουργία μη κυβερνητικών οργανώσεων στη χώρα αυτή. Παρακαλώ, κυρία Μπρεπούλς. Δεν απατώμε, αλλά πρέπει να πω προηγουμένως κάτι, ο πρόεδρος. Και αυτό είναι ότι θα δούμε πρώτα την ερώτηση που έχει να κάνει με τους σπόρους για την Κούβα. Και μετά θα πάμε στην ερώτηση της κυρίας Μπίπουλς. Ευχαριστώ. Ε, εκ μέρους της κυρίας Αντρικέτη θέλω και εγώ να ρωτήσω κάτι. Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που αντικαθιστά ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία. Ξέρουμε ότι πρικοδοτείται με ένα σημαντικό προϋπολογισμό. Από σήμερα, το μέσο αυτό ε, χρησιμοποιείται σε πάνω από 100 χώρες, ε, και αναρωτιόμαστε γιατί δεν καλύπτεται εκεί η Κούβα από αυτό το μέσο, εκεί όπου επιδόσεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, δεν πάει καθόλου καλά. Θα μπορούσαμε να πιέσουμε ίσως ε, βλέποντας ποια τελικά προγράμματα θα χρηματοδοτήσουμε και ποια όχι με αυτό το μέσο. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σας. Όσον αφορά την ερώτησή σας αυτή, εγώ θα έλεγα ότι πριν από το 2008, όπου είχαμε ξανά συνεργασία με την ε, Κούβα, τότε είχαμε διάφορα προγράμματα που χρηματοδοτούσαμε μέσω του μέσου αυτού για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, επικεντρωνόμενοι κυρίως σε προγράμματα κοινωνικής συνοχής. Πιο πρόσφατα όμως, ε, την ε, στήριξή μας τη δώσαμε και σε άλλα προγράμματα που είχαμε νωρίτερα μέσω μη κυβερνητικών ε, παραγόντων. Και από τότε που ξανάρχισε η συνεργασία μας, το 2008, έχουμε επηρεάσει πολύ περισσότερο τα πράγματα με διάφορα προγράμματα με 3 εκατομμύρια για τέτοιου είδους προγράμματα. Πριν ήταν 300.000. Η βασική ιδέα, Πρόεδρε, είναι η εξής. Υπάρχει ένας ανοιχτός τρόπος με τον οποίο γίνονται τα προγράμματα αυτά. Λαμβάνουμε υπόψη μας ότι στην Κούβα η κυβέρνηση δεν βλέπει τις δραστηριότητες αυτές σαν να συνάδουν με την υπάρχουσα νομοθεσία. Τα προγράμματα, δηλαδή αυτά, όταν τίθεται σε εφαρμογή, θέτουν σε κίνδυνο αυτούς που τα εφαρμόζουν. Και το ξέρουμε αυτό, το έχουμε διαπιστώσει. Και από τις Ηνωμένε Πολιτείες ξέρουμε ότι ένας δικός τους ε, συνελήφθη και καταδικάστηκε σε μακροχρόνιο φυλάκιση. Κάτι το οποίο βέβαια είναι μεγάλο πρόβλημα και για τον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά και για τα προγράμματα και για όλη την διαδικασία στήριξης των ΗΠΑ. Τώρα η δικιά μας υπηρεσία εξωτερικής δράσης έχει δεσμευτεί να στηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα πολιτικά δικαιώματα στην Κούβα. Γι' αυτό και συνεχίζουμε πολιτικό διάλογο με την Κούβα και πιστεύουμε ότι έχουμε προχωρήσει μέσω αυτού του πολιτικού διαλόγου, έχουμε κάποια αποτελέσματα. Παρόλο που δεν μπορεί φυσικά να πει κανείς ότι ο πολιτικός διάλογος με την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί και το, τη μόνη αιτία, το μόνο λόγο που αλλάζουν τα πράγματα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κούβα, αλλά παρόλα αυτά ο πολιτικός μας διάλογος έχει συνεισφέρει και αυτός στην πρόσφερη απελευθέρωση πολιτικών κρατούμενων στην Κούβα. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία και την έκθεσή της δεν υπάρχουν πια πολιτικοί κρατούμενοι στην Κούβα. Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ σημαντική. Και πιστεύω ότι ο πολιτικός διάλογος και η πολιτική δέσμευση που ακολουθούμε υπέρ της πολιτικής μας αυτής και της πολιτικής των κρατών μελών έχει αποφέρει καρπούς. Όπως είπα και νωρίτερα λοιπόν, τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στο κέντρο των σχέσεών μας με την Κούβα και θα συνεχίσουμε στην ίδια αυτή γραμμή με πολιτικό διάλογο με τη χώρα αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι. Κύριος Ντάνσκης έχει κάτι να συμπληρώσει. Ναι, ευχαριστώ. Θα περάσουμε τώρα, λέει ο Πρόεδρος, στην ερώτηση της κυρίας Μπρίσπολ. Πρόκειται για τις νομοθετικές ρυθμίσεις τις οποίες έχει προχωρήσει το Ισραήλ και που αποτελούν εμπόδιο στη λειτουργία των μη κυβερνητικών οργανώσεων στη χώρα αυτή. Κύριε Πρέπουλς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, πράγματι πρόκειται για την κατάσταση των μη κυβερνητικών οργανώσεων στο Ισραήλ. Και δεν είναι η πρώτη φορά, νομίζω, που εξετάζουμε το ζήτημα αυτό εδώ, στην Επιτροπή μας αυτή και γενικότερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλές φορές μέχρι τώρα έχουμε εκφράσει την ανησυχία μας με ψήφισμα, για παράδειγμα που έχουμε εγκρίνει και όπου προτείναμε κάτι σχετικά με την ε, νομοθεσία από την ΚΝΕΣΕΤ που πριν από λίγες εβδομάδες ψήφισε μια ρύθμιση με την οποία περιορίζεται η λειτουργία μη κυβερνητικών οργανώσεων. Έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση που μπορούν να έχουν ε, αυτές από το εξωτερικό, αλλά και με άλλα θέματα. Τα οποία σίγουρα μπορούν να επηρεάσουν πάρα πολύ προς το χειρότερο τη δουλειά που μπορούν να κάνουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις στο Ισραήλ. Ξέρω ότι οι προτάσεις δεν έχουν περάσει συνολικά από την ΚΝΕΣΕΤ γιατί συνεχίζεται η συζήτηση στην ε, ΚΝΕΣΕΤ μεταξύ των διαφόρων πολιτικών πλευρών. Παρ' αυτά οι προτάσεις υπάρχουν και έχουν εγκριθεί στην αρμόδια επιτροπή τους. Οπότε το πιο πιθανό είναι να περάσουν και στην Ολομέλεια της Κνασέτ. Και θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο, αλλά μου έχουν απαντήσει γραπτά έτσι καλώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε θα αρκεστώ σε αυτό. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε. Κυρία Μπρέπουλς. Ο κύριος Γαμπρίτσης, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, Θέλω να υπογραμμίσω ότι πράγματι μόλις ακούσαμε για το νομοσχέδιο αυτό στο οποίο αναφερθήκατε και εμείς ε, ανησυχήσαμε γιατί όντως ο τρόπος και το περιεχόμενο του νομοσχεδίου δεν είναι κάτι το οποίο μας αρέσει να έχουμε μπροστά μας όταν ε, έχουμε διμερείς σχέσεις με κάποια χώρα. Γι' αυτό και δραστηριοποιηθήκαμε αμέσως και μέσω του πρέσβη μας εκεί τόπου και εδώ μέσω της πρεσβείας του Ισραήλ σε μας και η εξωτερική υπηρεσία αλλά και τα κράτη-μέλη δραστηριοποιηθήκαμε. Διότι όλοι συμμεριζόμαστε, αποκοινούμε το Συμβούλιο την ανησυχία αυτή. Δεύτερον, θέλω να πιστεύω ότι το πάγωμα της πρωτοβουλίας αυτής αποτελεί καρπό των προσπαθειών που κάναμε εμείς και του μηνύματος που του στείλαμε. Βέβαια, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, δεν είναι επειδή προς το παρόν έχει παγώσει το θέμα ότι δεν θα προωθηθεί ίσως με διαφορετικό τρόπο. Γι' αυτό και δεν πρέπει να ολιγορούμε και πρέπει στον πολιτικό διάλογο που θα έχουμε και την επόμενη εβδομάδα με το Ισραήλ να φροντίσουμε να το συζητήσουμε. Πρέπει να επαγρυπνούμε. Θα ήθελα όμως, αν μου επιτρέπετε, να κάνω και δύο άλλες παρατηρήσεις, παρακαλώ, σχετικά με την αντίδρασή μας. Πρώτον, σχετικά με την αναγκαιότητα που υπάρχει να συνεχίζουμε κράτη, μέλη, Συμβούλιο, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, Επιτροπή, Κοινοβούλιο, να συνεχίζουμε. Βλέπετε, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια συνάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με εκπροσώπους της ΚΝΕΣΕΤ που είχαν έρθει εδώ στο Κοινοβούλιο και θίξαμε το θέμα αυτό. Ήταν ξεκάθαρο ότι οι φίλοι μας εκπρόσωποι της Κνεσέτα στη συνεδρίαση αυτή και αυτοί εξέφρασαν την ανησυχία τους. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, και μέσα στο Ισραήλ γίνεται συζήτηση για αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει συμφωνία δηλαδή. Πώς να το πω, με άλλα λόγια, πρέπει να υποφεληθούμε από τις διμερείς σχέσεις που έχουμε για να τροφοδοτούμε και άλλο τη συζήτηση στο εσωτερικό του Ισραήλ. Αυτό δηλαδή είναι ένας δρόμος, ένα μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας για να πιέσουμε, να επηρεάσουμε ώστε να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια και πραγματική εταιρική σχέση. Γιατί δεν είναι μόνο να πούμε, ξέρετε, είναι ανισχυτικό ο νόμος αυτός που κινδυνεύει να περάσει στο Ισραήλ, όχι, αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις κοινέ αξίες μας, να τις βάλουμε στο τραπέζι κατά τον πολιτικό διάλογο και σε συνεργασία και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, τροφοδοτούμε όσο γίνεται πιο θετικά και επικοδομητικά τη συζήτηση που ήδη γίνεται μέσα στο Ισραήλ. Και δεύτερον, δεύτερη παρατήρηση που ήθελα να κάνω, Όταν έχουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, συχνά από πίσω υπάρχουν κάποιες αιτίες, κάποιοι λόγοι, κάποιοι στόχοι. Θα πρέπει και εμείς να προσπαθούμε να καταλαβαίνουμε Ποιος είναι ο λόγος που οδηγεί σε μια τέτοια πρόταση. Κάποιους μπορεί να τους καταλαβαίνουμε, κάποιους όχι, με κάποιους μπορεί να συμμεριζόμαστε, κάποιους όχι, εξάλλου τους αναφέρετε κι εσείς με την ερώτησή σας. Αλλά γι' αυτό ίσως θα πρέπει να παρακολουθούμε γενικότερα τις δράσεις των μη κυβερνητικών οργανώσεων γιατί για χίλιες ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις που λειτουργούν καλά μπορεί να υπάρχει και μία η οποία δεν εντάσσεται απαραίτητα στο πνεύμα καλής λειτουργίας όπως θα περιμέναμε από μια μη κυβερνητική οργάνωση. Όπως και να έχει το πράγμα, εμείς εξακολουθούμε να χρηματοδοτούμε είτε διμερώς είτε σε περιφερειακό επίπεδο διάφορα προγράμματα εμείς δεν χρηματοδοτούμε μη κυβερνητικέ οργανώσεις, αλλά προγράμματα άπαξ και ε, έχουμε κρίνει ότι είναι καλά τα προγράμματα αυτά. Η χρηματοδότηση της κοινωνίας των πολιτών τόσο στο Ισραήλ όσο και σε ολόκληρη την περιοχή είναι κάτι πολύ σημαντικό και για μας συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Γκαμπρίτσι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάτι πρακτικό για το τέταρτο ερώτημα που έθεσε η κυρία Μπρέμπολς για τις επιπτώσεις που θα, είχαν, είχε η νομοθεσία αυτή στον προπολογισμό των μη κυβερνητικών. Ε, εμείς δεν θα μειώσουμε το χρηματοδότηση, αλλά έχουμε δώσει και άλλα 500.000 ευρώ για το 2012 για να υπάρξει υποβολή προτάσεων, τις οποίες βεβαίως θα διαχειριστεί η αντιπροσωπεία μας στο Τελαβίβ. Μετά από συνεννόηση με τα κεντρικά θα μπορέσει να ληφθεί απόφαση για το πού θα πρέπει να πάνε τελικά αυτά τα κονδύλια, τα οποία μπορούν να είναι είτε ως ενίσχυση της τοπικής ε, κοινωνίας των πολιτών, είτε για δράσεις ε, που σχετίζονται με την ελευθερία. Ε, υπάρχει βέβαια και ένα θέμα φορολόγησης ε, δύναμη της ε, νομοθεσίας του Ισραήλ που μπορεί να επηρεάσει τα προγράμματα που εμπίπτουν στο EMPI και τα ποσά αυτά της φορολόγησης δεν μπορούν να κτηθούν από, με άλλο τρόπο. Η νομοθεσία προς το παρόν δεν το επιτρέπει αυτό, οπότε μάλλον θα πρέπει να το δούμε σε πιο γενικούς όρους στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω πώς θέλετε, κυρία Μπρέπολς, και πάλι το λόγο. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Ε... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ όλους όσοι απάντησαν και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την εξωτερική δράση. Τους ευχαριστώ όλους για τις πληροφορίες τους. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό η πρωτοβουλία αυτή να μην μείνει έτσι. Πρέπει να παρακολουθούμε πολύ καλά το τι γίνεται. Υπάρχει κάποιος κίνδυνος εδώ. Ε, ξέρετε πώς έχει κατάσταση με τη βία στην περιοχή, οπότε τέτοιες ε, ε, πρωτοβουλίες από μη κυβερνητικέ οργανώσεις είναι σημαντικές και καταλαβαίνετε πως ε, η νομοθετική αυτή πρόταση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον τρόπο λειτουργίας των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Καλό θα ήταν να μην προχωρήσει άλλο η πρωτοβουλία αυτή Καταλαβαίνετε και μόνο που υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία θα το σκεφτούν πολύ να προσλάβουν κάποιον όπως είχε γίνει με τον κύριο Κόλμα, θα θυμόσαστε. Πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να αντιδράμε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν συμφωνεί με αυτή την πρωτοβουλία Εξάλλου έχουμε και την ε, δήλωση του ΙΕ για αυτό το θέμα. Ελπίζω ότι θα το χρησιμοποιήσετε και αυτό και ότι θα πετύχετε τέτοιου είδους νομοθετικές πρωτοβουλίες να αποφεύγονται στο μέλλον και να μην είναι δυνατόν να προχωράνε. Ευχαριστώ πάντως για τις προσπάθειές σας. Ο Πρόεδρος. Θέλετε να απαντήσετε, κύριε Γκαμπριτσί. Απλώ κάτι να επενθυμίσω ακριβώ, όπω είπαμε για την επόμενη εβδομάδα, πρόκειται να έχουμε πολιτικό διάλογο με το Ισραήλ και οπότε το θέμα αυτό θα συνεχιστεί να συζητείτε. Και στη διάθεσή σα να συνεχίσω να σα ενημερώνω όσον αφορά τι ε, μέλουσε εξελίξει. Είναι κάτι το οποίο δεν θα λυθεί από τη μία μέρα στην άλλη, θα πρέπει να το παρακολουθούμε να υπάρχει διαφάνεια όπως είπα και έτσι να μπορέσουμε να έχουμε κάποια τα αποτελέσματα. Ποια σας πω τι θα γίνει με την συνάντηση αυτή με τους Ισραηλινούς την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα πάμε στο επόμενο θέμα. Άννα Γκόμες. Αλλά θα μας μιλήσει για αυτό το θέμα ο κύριος Πρόντι, έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Η συνάδελφος ακόμα δυστυχώς δεν μπορεί να παραστεί σήμερα εδώ και μου ζήτησε εγώ να σας παρουσιάσω το θέμα της. Βεβαίως, εννοείται ότι συμφωνώ 100% με τις θέσεις της Πρόκειται για αυτή την ε, προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το Αφγανιστάν για ε, την προστασία των γυναικών κατά της καταπάτησης των ε, δικαιωμάτων τους είναι σαφές ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και σχετίζεται άμεσα με το δικό μας έργο. είναι μια ταινία, ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο ολοκληρώθηκε το Μάρτιο. Χρηματοδοτήθηκε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν όμως ολοκληρώθηκε το ντοκιμαντέρ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλησε να αποσύρει την υποστήριξή της για να προστατεύσει τις γυναίκες που εμφανίζονται σε αυτήν την ταινία, σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Οι αναγκόμενες και υποφαινόμενες θα θέλαμε να απευθυνθούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην εξωτερική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δούμε τι θα γίνει ε, Πώς έχει η κατάσταση για αυτή την ε, μάλλον πολιτική απόφαση. Ήταν πολιτική απόφαση, δεν είναι πρόκειτο για προσπάθεια προστασίας των ε, γυναικών που εμφανίζονται στην ταινία. Πάντως, δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις προσπάθειές μας, να επισημαίνουμε ένα πάρα πολύ αμφίβολης διαφάνειας σύστημα το οποίο επικρατεί στο Αφγανιστάν θα πρέπει και νομοθετική εξουσία και δικαστική να κάνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις. Αυτά με γενικές, σε γενικές γραμμές. Έτσι έχει το θέμα αυτό στο Αφγανιστάν. Πρόκειται για μια κατάσταση επομένως η οποία μας προβληματίζει πολύ. Και θα πρέπει επομένως να δούμε πώς θα γίνονται σεβαστά τα ατομικά δικαιώματα. Γι' αυτό και θέλουμε και στην Ευρωπαϊκή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απευθυνθούμε και να του ρωτήσουμε σχετικά. Ευχαριστούμε, λίγο Πρόεδρος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλετε να λάβετε το λόγο μας εξηγήσετε τι συνέβη. Good morning, uh, Καλημέρα σας. Να σας ευχαριστήσω για την ε, ευκαιρία που μου δίνετε να εξηγήσω λίγο το τι συνέβη. Να σας ε, διαβεβαιώσω ότι το σημείο αυτό, το θέμα αυτό μας απασχολεί και μας και βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα μας ακριβώς για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αφγανιστάν. Να σας εξηγήσω όμως λίγο τι έχει γίνει. Όταν ε, η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής ε, ε, Ένωσης συζητούσε το θέμα της χρηματοδότησης πέρσι, είχαμε σκοπό να ρίξουμε περισσότερο φως στα θέματα των συγκατάσταση μάλλον που επικρατεί στο Αφγανιστάν με τις γυναίκες. Είναι πολύ δύσκολο, πολύ ευαίσθητο το θέμα αυτό και Κυρίω το θέμα σε, τον, η κατάσταση των γυναικών σε περιπτώσει εντάσεων. Προσπαθήσαμε λοιπόν να το δούμε το θέμα αυτό, γιατί ακριβώ ε, έχει να κάνει και με τα ανθρώπινα δικαιώματα και με τη δικαιοσύνη που αποτελούν τα σημεία κλειδιά στις σχέσεις μας με το Αφγανιστάν. Αυτό έχει να κάνει και με την αναπτυξιακή ε, συνεργασία ε, και με την συνεργασία μας γενικώ με την κοινωνία των πολιτών και τους οργανισμούς, τις οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως έχουμε τώρα την τελική εκδοχή του, της, ε, του κειμένου, έχουμε πάρα πολλές ανησυχίες. Γιατί αναφέρει τα βασικά προβλήματα του σοφρονιστικού συστήματος στο Αφγανιστάν, αλλά το πρόβλημα είναι ότι το κάνει με τέτοιο τρόπο ε, που να αποκαλύπτει απόλυτα την ταυτότητα των γυναικών. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας εξηγήσω ότι σε ένα τέτοιο, στα πλαίσια ας πούμε, της κοινωνίας το να, της Αφγανικής το να ε, παρουσιαστεί, να φανερωθεί η ταυτότητά τους, η ταυτότητά τους μπορεί να είναι απειλή, μπορεί να αποτελεί και απειλή για τη ζωή τους. Με βάση λοιπόν όλα αυτά, η αντιπροσωπεία στο Αφγανιστάν της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ότι το φιλμ αυτό δεν θα μπορούσε να ε, προβληθεί στην παρούσα εκδοχή του επαναλαμβάνω, έτσι όπως είναι τώρα. Για να είναι λοιπόν τα πράγματα σαφή, η χώρα αυτή είναι μια χώρα όπου ένα θύμα βιασμού είναι ντροπή, αποτελεί ντροπή για την, κοινωνία, για την οικογένειά του. Συγγνώμη. Και η, φόνοι φόνη τιμή, τα εγκλήματα τιμή είναι πολύ συχνά. Οι γυναίκε λοιπόν υποφέρουν πολύ, ούτω ή άλλω, υπό τι παρούσε συνθήκε. Η απόφαση λοιπόν που ελήφθη ήταν να μην προβληθεί το φιλμ αυτό, η ταινία, στην ε, παρούσα της μορφή και ε, αυτή η απόφαση βασίστηκε μόνο στην ε, προσπάθεια προστασίας των γυναικών. Δεν ήταν εύκολο να ληφθεί η απόφαση αυτή. κάναμε πολλές διαβουλεύσεις με την Κομισιόν, με την, με τον, με την EAS, με την αντιπροσωπεία μας και με τους εμπρογνώμονες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με, ήρθαμε σε επαφή με μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Έγιναν λοιπόν πολλές συζητήσεις πριν ληφθεί τελική απόφαση από την αντιπροσωπεία. Αυτό τώρα που μένει εμείς να κάνουμε είναι οι γυναίκες που μέσα στην, ε, που παρουσιάζονται μέσα στην ταινία ε, να σεβαστούμε την επιθυμία που εξέφρασαν ότι δεν θέλουν και αυτές να παρουσιαστεί, να προβληθεί η ταινία αυτή. Το έχουν καταστήσει απόλυτα σαφές. Αν τώρα προβληθεί η ταινία αυτή, Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε, δεν μπορούμε να αποφύγουμε με κανέναν τρόπο να μπει το, η ταινία αυτή στο ίντερνετ και να παρουσιαστεί παντού. Και ήθελα να πω ότι έχουν γίνει και με τους παραγωγούς της ταινίας συζητήσεις και τους έχουμε ζητήσει να ε, κρύψουν την ε, ε, ταυτότητα των γυναικών, να θολώσουν τα πρόσωπά τους στο, μέσα στην ταινία, να αλλάξουν λίγο τα πράγματα, τις, τα όσα αναφέρονται δηλαδή, έτσι ώστε να μην μπορούν να αναγνωριστούν. Δυστυχώς ο παραγωγός της δεν το έχει κάνει, δεν συμφώνησε σε κάτι τέτοιο. Τώρα για το δεύτερο τμήμα της ερώτησής σας, συμφωνώ απόλυτα ότι όντως πρέπει να δούμε το θέμα της, ε, ε, του σοφρονιστικού συστήματος ε, και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αφγανιστάν, ειδικά την, την, κράτηση των, την κατάσταση των γυναικών κρατουμένων. Γνωρίζουμε ότι το κράτος δικαίου του, δικαίου του Αφγανιστάν είναι πολύ αδύναμο και οι γυναίκες και τα παιδιά είναι οι πιο ευπαθείς ομάδες από όλη την κοινωνία. Όχι μόνο σε διαφορά την πρόσβαση σε νόμο, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό έχουμε κάνει, έχουμε θέσει ως ε, προτεραιότητα των προγραμμάτων μας την μεταρρύθμιση του σοφρονιστικού συστήματος με προγράμματα που θα ενισχύσουν τη γνώση για τα συνταγματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα των γυναικών στο Ισλάμ, ε, προσφορά νομικών υπηρεσιών ε, σε γυναίκες που έχουν υποφέρει από ενδοοικογενειακή βία έτσι ώστε να έχουμε ένα ευρύ φάσμα προ... προστασίας της... προς τις γυναίκες του Αφγανιστάν. Η βελτίωση της ε, κατάστασης βεβαίως στο Αφγανιστάν είναι μια διαδικασία μακρά. Δεν θα έρθει από εν μια ανοιχτή η αλλαγή. Πρέπει λοιπόν όλοι να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση μέσω διαφορετικών όμως ε, δομών συμπεριλαμβανομένου και του διαλόγου με τις αφγανικές αρχές. Δεν ε, κρυβόμαστε, προσπαθούμε να θίγουμε πάντα τα θέματα αυτά με τους, αφγανικές αρχές. Και επίσης η Κομισιόν έχει συμφωνήσει ότι όντως ε, πρέπει να υπάρξει ε, καταγραφή των ε, μη δικαίων πρακτικών Και βεβαίω το να μην προβληθεί η ταινία αυτή δεν έχει να κάνει με πολιτικέ πτυχέ. Δηλαδή δεν θα επηρεάσει το να μην προβληθεί η ταινία τι σχέσει που έχουμε με τι αφγανικέ αρχέ ή τη δουλειά που έχουμε κάνει. Έχει να κάνει μόνο με τη βασική υποχρέωση και ευθύνη να μην ε, παρουσιάζονται οι γυναίκες αυτές, να μην αναγνωρίζονται οι γυναίκες που παίρνουν μέρος ε, σε αυτή την ταινία, έτσι ώστε να μπορούν να αποφευθούν οι συνέπειες που μπορεί να είναι και απειλητικέ για τη δική τους τη ζωή ή ακόμη και να ε, ε χειροτερεύσουν ακόμη περισσότερο τις, τα μαρτύρια που υποφέρουν τώρα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ωραία, λοιπόν, ακούσαμε τι μας είπε η Κομισιόν. Κύριε Πρόεδρε, θέλετε το λόγο και πάλι. Ε, ε. Ναι, ναι, Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Αν ε, η κατάσταση αυτή όντως είναι ισχύει, τότε θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί ίσως και θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες ε, εγγυήσεις έτσι ώστε από την αρχή να μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια αυτών των ανθρώπων. Ό,τι και να γίνει φαίνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί το ποσό για την παραγωγή αυτής της ταινία. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να ξαναγίνει από την αρχή. Συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρχει το ανώτατο επίπεδο ασφάλειας για τις γυναίκες αυτές που ήδη έχουν υποφέρει τρομερά. Το πρόβλημα ουσιαστικά, αν έχω καταλάβει καλά, είναι ότι αυτό το, αυτή η ταινία τελικά δεν θα χρησιμοποιηθεί καθόλου. Ευχαριστώ για το ερώτημά σας. Αυτή η ταινία μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Και όπως είπα, η απόφαση να μην επιτρέψουμε την προβολή της, έτσι όπως είναι, δεν ήταν εύκολη απόφαση. Γνωρίζουμε ότι από τη μια η παρουσίαση της, των, της κατάστασης των γυναικών σε κράτηση μπορεί να βοηθήσει γενικώ τις γυναίκες στο Αφγανιστάν και οποιαδήποτε άλλη γυναίκα βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση. Αλλά απ' την άλλη κατανοούμε ότι δεν μπορούμε να εκθέσουμε αυτές τις γυναίκες. Μπορεί αυτό να αξιολογηθεί βεβαίως μόνο όταν... Αυτό μπορούσε να αξιολογηθεί μόνο όταν είδαμε την τελική εκδοχή της ε, ταινία. Εξεκολουθώ να ελπίζω ότι το, η ταινία αυτή θα μπορέσει να... να αναπροσαρμοστεί εν πάση περιπτώσει και να, την, και να προβληθεί. Ευχαριστώ. Είμαι από την Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά. Ήθελα να απαντήσω κι εγώ. Βεβαίως δεν ε, αποφεύγουμε να θίξουμε τα θέματα αυτά σε κάθε περίπτωση στις ε, ε, αφγανικές αρχές. Το κάνουμε και ιδιωτικά μέσω ας πούμε των επικεφαλής της, των αποστολών ή της αντιπροσωπείας αλλά το κάνουμε και όταν αυτό είναι σωστό δημοσίως ας πούμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα που ήταν όντως πολύ σημαντικό. Έχουν υπάρξει πολλές συζητήσει ε, για, ένα νέο, για μια νέα νομοθεσία για το άσυλο. Ε, αυτή η νομοθεσία ήταν σωστή και ήταν μια καλή προσπάθεια από τις αφγανικές αρχές να ρυθμίσουν το ευρύ αυτό θέμα του ασύλου. Αλλά κάποια τμήματα αυτής της νομοθεσίας θα ήταν πραγματικά πολύ παρεμβατικά και παρόμοια με το θέμα που συζητούμε εδώ, θα έθεταν σε κίνδυνο την, την ζωή των γυναικών. Και αν το είχε επιτρέψει αυτό η διεθνής κοινότητα, θα είχε μεγάλο, μεγάλο θα υπήρχαν πολλές, περιπτώσεις μετά από εκεί και πέρα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και η Πατή Εκπρόσωπος εξέδωσε λοιπόν μία δήλωση Αποκινούμε άλλα μέλη της, διεθνής, της κοινότητας για την, για την αναθεωρημένη νομοθεσία α, για το άσυλο η οποία τώρα, μετά από παρεμβάσεις, είναι ε, αποδεκτή από τις, από τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της χώρας. Οπότε, να, ας πούμε, ένας τρόπος για να λύσουμε τέτοιου είδους ζητήματα. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Οπότε τώρα έχουμε ολοκληρώσει τις ε, ερωτήσεις που έπρεπε να απορριφθούν σήμερα. Τώρα το επόμενο σημείο στις 10 η ώρα. Άρα έχουμε μισή ώρα διάλειμμα. Κυρίε Κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε. Θα επικεντρωθούμε στην ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Δυτική Παππούα και την Ινδονησία. Συνεχίζω στα πολωνικά. Καλώς ήρθατε λοιπόν και πάλι. Έχουμε μία ακρόαση για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Νότιο Ανατολική Ασία. It's okay. Have you translation? Yes, yes. Uh, serdecznie witam Państwa w tej części posiedzenia. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Το ξαναλέω γιατί υπήρξε ένα πρόβλημα έχουμε μία ακρόαση για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Νότιο-Ανατολική Ασία. και κυρίως στην Δυτική Παπούα και την Ινδονησία. Προς το παρόν, στην Ινδονησία η Ινδονησία μάλλον, ε, αποτελεί μια πιο ανοιχτή, πιο ανεκτική κοινωνία. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι όλες αυτές οι αλλαγές, οι θετικές αλλαγές στην Ινδονησία μπορεί να, μπορούν να οδηγήσουν στο να γίνει υπόδειγμα η, ε, ε, Ινδονησία. Παρ' αυτά, είναι, αδύναμες, είναι αδύναμοι οι θεσμοί της Ινδονησίας. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα διαφθοράς. Και πέρα από αυτό... Υπάρχουν προβλήματα με, την, με τον πληθυσμό που είναι ανησυχητικά. Η Παπούα είναι το νότιο τμήμα της ε, Νέας Γουινέας, αποτελεί τμήμα της, ε, ε, της, της Ινδονησίας, της Ινδονησίας από το 1969. Έχουν υπάρξει πάρα, πολλές, πάρα πολλά πραξικοπήματα, έχουν υπάρξει πολλές φορές προσπάθειες με, με στρατιωτικά μέσα να υπάρξει ε, η διακυβέρνηση της χώρας αυτής. Βεβαίως έχει υπάρξει τεράστια αντίδραση από τους ε, αυτόχθονες και η προσέγγιση αυτή έχει οδηγήσει στο να υπάρχουν πάντα παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δυτική Παπούα. Έχουμε λοιπόν πολλούς προσκεκλημένους σήμερα που γνωρίζουν πολύ καλά τα πράγματα στη συγκεκριμένη αυτή περιοχή. Ο καθένας θα μιλήσει περίπου 10 λεπτά, έτσι ώστε να έχουμε την δυνατότητα να θέσουμε και ερωτήματα. Και βεβαίως οι προσυκλημένοι μας θα απαντήσουν στις ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών. Να πω επίσης ότι ε, έχουμε και προσκεκλημένο από την Ολλανδία. Δεν ξέρω βεβαίω αν είναι ήδη εδώ. Μάλλον όχι, από ό,τι βλέπω. Θα χαρούμε βεβαίω να τον ε, καλωσορίσουμε μόλι φτάσει. Οπότε, να ακούσουμε πρώτα τον ε, κύριο Μπάρμπερ, ο οποίος είναι συντονιστής της ΤΑΠΟΛ, των ε, πολιτικών κρατουμένων δηλαδή, της οργάνωσης που ασχολείται με τους πολιτικούς ε, κρατούμενους. Ασχολείται λοιπόν η οργάνωση αυτή, η ΤΑΠΟΛ, με την ε, εγκαθίδρυση της δημοκρατίας και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κύριος Μπάρμπερ λοιπόν είναι ο συντονιστής της ΤΑΠΟΛ, ο οποίος θα μας παρουσιάσει την κατάσταση στη Δυτική Παππούα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ και τα μέλη της Υποεπιτροπής σας που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για την Δυτική Παππούα σήμερα. Θα ήθελα να μοιράσω την παρουσίασή μου σε τρία μέρη. Το πρώτο θα σας δώσει κάποιες πληροφορίες για τη Δυτική Παππούα. Το δεύτερο θα καλύψει πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις και το τρίτο θα αναφέρει τα προβλήματα που υπάρχουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα προτείνει συγκεκριμένες επικοδομητικές λύσεις για να δημιουργηθεί ο χώρος που χρειάζεται έτσι ώστε να υπάρξει ειρηνική λύση της διαμάχης που υπάρχει στη Δυτική Παππούα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σωστή η χρονική στιγμή που μιλούμε για το θέμα της Δυτικής Παππούα γιατί τα θέματα και οι εντάσει που προκύπτουν ε, από την, στην χώρα αυτή θα είναι πολύ σημαντικές. Ε, την Πέμπτη, πριν από πολλά χρόνια, το 1961, ε, στα πλαίσια της διαδικασίας της Ολλανδικής διακυβέρνησης που θα οδηγούσε σε αυτοδιάθεση της Παππούα, βασικά σύμβολα της, της εθνικότητας της Παππούα, όπως ας πούμε η σημαία και ο εθνικός ύμνος, ε, υιοθετήθηκαν επισήμως από τους εκπροσώπους της Παπούα με την παρουσία και ε, Ολλανδών αξιωματούχων. Από τότε, η 1η Δεκεμβρίου εορτάζεται από τους αυτόχθονες ως η εθνική τους ημέρα, ημέρα ή ημέρα της ανεξαρτησίας. Ε, η φετινή επέτειος είναι πολύ σημαντική, γιατί είναι η πεντηκοστή επέτειος και έρχεται σε μια χρονική στιγμή ιδιαίτερης πολιτικής αστάθειας και βίας στην ε, περιοχή. Δυστυχώς, ε, ο, ο Πάτερ Τιμπέι, ε, που απολαμβάνει μεγάλου σεβασμού και ήταν μέλος της του δικτύου για την ειρήνη δυστυχώς ακύρωσε την παρουσία του εδώ γιατί πραγματικά ανησυχούσε πάρα πολύ και την κατάσταση στη χώρα. Έχει στείλει όμως ένα μήνυμα το οποίο θα το διαβάσω μετά τη δική μου παρουσίαση. Η, ε, η ανεξάρτητη διακυβέρνηση στην Παππούα δεν ε, ευδοκίμησε ποτέ, αλλά υπάρχει αυτή η πολύ περίπλοκη διαδικασία της πράξης της ελεύθερης επιλογής ε, που οδήγησε στην προσάρτηση στην Ινδονησία το 1969. Από τότε οι αρχές της Ινδονησίας έχουν ε, ε, επιλέξει μια πολύ στρατιωτική και αυστηρή προσέγγιση για να έχουν την κυριαρχία στην περιοχή ε, Βεβαίω, ε, υπάρχει μεγάλη αντίθεση από την Τζακάρτα για τα δικαιώματα των ε, πολιτών τη Παππούας. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν μια μεγάλη ένταση κατά της Τζακάρτα, κάτι που τροφοδοτεί ακόμη περισσότερο την διαμάχη αυτή. Βεβαίω, έχουν υπάρξει πολλές περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρόλο που έχουν ε, ε, εγκαταληφθεί οι φυσικοί πόροι και έχουν αποτελέσει το μεγαλύτερο φορολογούμενο της Ινδονησίας, ε, η Δυτική Παππούα είναι μία από τις πιο φτωχές περιοχές της Ινδονησίας ό,τι αφορά τα επίπεδα φτώχειας και τους δείκτες ανθρώπινης ανάπτυξης μεγάλες ε, χώρες, ε, δασικές, μεγάλες περιοχές ε, δασικές στοχεύονται για την παραγωγή τροφίμων που βεβαίως αυτό έχει μεγάλες επιπτώσεις και για τους αυτόχθονες πληθυσμούς και για το περιβάλλον. Μετανάστες από άλλα κομμάτια, της, από άλλα μέρη της Ινδονησίας αποτελούν την, το βασικό πληθυσμό και δοκιμούν στην οικονομία θα, θα αποτελέσουν ε, συνολικά την πλειοψηφία έναντι των πολιτών της Παππούα. Και βρίσκονται λοιπόν οι πολίτες της Παππούα, οι αυτόχθονες, υπό μεγάλη απειλή. Ενώ ε, η Ινδονησία έχει κάνει μεγάλη πρόοδο στη, μεταφορά της, στη μετάβαση της ε, προς την ειρηνία από το 1998, οι, πληθυσμοί της Παππούα δεν έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία αυτή η ειδική αυτονομία που ε, δημιουργήθηκε το 2001 έχει απορριφθεί από, την, ε, από τη συνέλευση των ε, αυτοχθόνων γιατί δεν βελτιώνει τα δικαιώματα και τις συνθήκες διαβίωσης. Τώρα γίνονται προσπάθειες από τους θρησκευτικούς ηγέτες για να δημιουργηθεί ένας διάλογος με την κυβέρνηση της Ινδονησίας έτσι ώστε να επιτευχθεί μια ειρηνική επίλυση της σύραξης αυτής. Νωρίτερα φέτος, ε, υπήρξε μια διάσκεψη ειρήνης το, την οποία ε, οργάνωσε το δίκτυο ειρήνης από τις 5 έως 7 του Ιούλη στην Τζαϊπούρα δημιούργησε και έδωσε κάποια θετικά μηνύματα για το ότι γίνεται κάποια πρόοδος έτσι ώστε να επιληθούν τα προβλήματα της Παππούα. Το αποτέλεσμα αυτής της διάσκεψης ειρήνης έδωσε το πλαίσιο για ένα διάλογο με την κυβέρνηση της Ινδονησίας και κάποιες ε, προσδοκίες για, την, ε, μια ειρηνική Παππούα με καλύτερους ε, δείκτες που θα λένε πως η Παππούα είναι μια ειρηνική χώρα. Παρ' όλα αυτά δεν υποστηρίζουν όλοι οι πολίτες την διαδικασία αυτή διαλόγου γιατί δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση της συντονισίας. Κάποιοι πιστεύουν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πιο άμεση προσέγγιση όπως ας πούμε ένα δημοψήφισμα στο μέλλον σε κάθε περίπτωση η διαδικασία από την διάσκεψη μάλλον αυτή της ειρήνης έχουν ενταθεί ε, οι σειράξει στην ε, Παππούα, έχουν υπάρξει συλλήψεις, κρατήσεις, ε, βίες αντιδράσεις. Σύμφωνα με, την, με το Contrast που είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση έχουν σκοτωθεί πάνω από 40 άτομα. Οπότε μιλούμε για μια νέα περίοδο καταστολής. Εν τω μεταξύ έχει υπάρξει μεγάλη αντίσταση στα ε, λιμάνι από, από εργαζόμενους που ζητούν καλύτερους ε, μισθούς. Ε, και βεβαίως έχουν παρέμβει πολλές φορές οι δυνάμεις ασφαλείας με το θάνατο 10 ατόμων μεταξύ των οποίων και πολίτες και εργαζόμενοι και αστυνομικοί. Οι πρόσφατες λοιπόν αυτές βίες αντιδράσεις στην Παππούα κατέληξαν στην, στη δολοφονία τριών ατόμων μετά από ένα κογκρέσο που έγινε στην Τζαϊπούρ ε, από τις 16 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Ο στρατός και οι ειδικέ δυνάμεις της Ινδονησίας ε, πυροβόλησαν πάρα πολλές φορές για να μπορέσουν να διαλύσουν το πλήθος και χτύπησαν τους συμμετέχοντες. Ε, οι δυνάμεις ασφαλείας έγιναν βίες μετά από, τους, μετά από τη συγκέντρωση των ε, ηγετών που είχαν συγκεντρωθεί εκεί ε, και μετά την έκδοση ε, μιας δήλωσης ανεξαρτησίας. Αυτή λοιπόν η κατάσταση δείχνει ότι έχει υπάρξει αποτυχία από την πλευρά των αρχών της Ινδονησίας να διαχειριστεί ως ισότιμους ή να αντιμετωπίσει ως ισότιμους τους πολίτες της Παπούας. Έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο, το UP4B, το οποίο ε, έχει στόχο αυτό ακριβώς, την, ε, να ακουστεί η φωνή των ε, κατοίκων της Παππού, έτσι ώστε να προετοιμαστεί ο δρόμος για τον διάλογο. Ε, παραμένουν βεβαίω πολύ σημαντικά ερωτήματα για το κατά πόσο η Τζακάρτα είναι διατεθειμένη να θέσει τέτοια θέματα κοινωνικά και πολιτικά και οικονομικά στην ατζέντα. Υπάρχουν τρία θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα ήθελα να αναφέρω. Το πρώτο είναι η στρατικοποίηση, το, τρίτο, το δεύτερο είναι η ε, ατιμορρησία και το τρίτο είναι η ελευθερία της έκφρασης. Σύμφωνα με πρόσφατους υπολογισμούς, το προσωπικό της Δυτικής Παππούα ε, είναι περίπου 50.000 στις στρατιωτικές δυνάμεις. Ε, και υπάρχουν σχέδια να αυξηθούν πολύ κατά την επόμενη δεκαετία τα νούμερα αυτά. Αυτό βεβαίως είναι τελείως δυσανάλογο και πολύ αντιπαραγωγικό. Οι στρατιωτικέ επιχειρήσεις ε, και η αυστηρή αυτή προσέγγιση ε, αποτελεί μεγάλη παραβίαση και απειλή προς τα δικαιώματα των πολίτων της Παππούα. Οι δυνάμει ασφαλεία θεωρούν ότι η πολιτική δραστηριότητα και, τα, και η υπεράσπιση των ε, δικαιωμάτων των πολιτών, των πολιτών της Παππούα έχει να κάνει με την διάθεση ανεξαρτητοποίησης αυτών και θα πρέπει να κατασταλεί. Υπάρχουν τεράστιοι περιορισμοί σε, έναντι εξωτερ, ε, αλλοδαπών ΜΜΕ και οργανισμών που σημαίνει ότι ε, ο έλεγχος και η παρακολούθηση των δράσεων των αστυνομικών δυνάμεων δεν μπορεί να γίνει καθόλου σε ό,τι αφορά το πρόβλημα αυτό, η Ινδονησία θα πρέπει να ενθαρρυνθεί για να δει το θέμα της πολιτικής, της στρατιωτικής και αστυνομικής της σε ό,τι αφορά την Παπούα, μειώνοντα την παρουσία του στρατού εκεί και επικεντρωνόμενη ε, περισσότερο στην ε, πολιτική προσέγγιση και όχι στην στρατιωτική για την επίλυση της διαμάχης αυτής. Επίσης θα πρέπει να επιτραπεί ε, άμεση ελεύθερη πρόσβαση στους πολίτες και ελευθερία εντός της Δυτικής Παππούας σε ό,τι αφορά την ε, πρόσβαση σε ανθρωπιστικές ε, ε, οργανώσεις καθώς και στα διεθνή ΜΜΕ. Οι πολίτε Παππούα τιμωρούνται για ειρηνικέ διαδικασίες, όπω α πούμε η, άρση της, η έπαρση τη σημαία. Σε αντίθεση με αυτό, οι αστυνομικέ δυνάμεις αναφέρουν ε, παρα, ε, που, που, πολλές, που παραβιάζουν πολλέ φορέ τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, εκφεύγουν οποιασδήποτε τιμωρία. Οχτώ αστυνομικοί οι οποίοι εμπλέκονται σε ε, μια καταστολή ενός κογκρέσου των ε, πολιτών της Παπούα απλώς ε, τους δόθηκε μια γραπτή προειδοποίηση. γιατί φαίνεται ότι ε, εγκαθιδρύεται μια ε, κατάσταση πλήρου τιμωρησία όπου ο καθένας μπορεί να κάνει οτιδήποτε και να μην τιμωρείται. Το Γενάρη του 2011 τρεις ε, στρατιώτες από στρατιωτικό δικαστήριο καταδικάστηκαν σε 8 με 10 μήνες φυλάκιση για την παράβαση εντολών. σε ό,τι αφορά τον δραματικό βασανισμό δύο ανθρώπων τον 2010. Ε, του 2010. Αυτό βεβαίω ε, έχει να κάνει με, τα, με τέτοια παρόμοια περιστατικά που συμβαίνουν εδώ και πολλά χρόνια. Η ατιμορρησία που υπάρχει λοιπόν είναι προφανή. Η κυβέρνηση τη Ινδονησία πρέπει να ενισχύσει τον ρόλο τη δική ε, Παππούα κάνοντα τι απαραίτητε έρευνε και διώξει των όσων συμμετείχαν σε, σε αυτές διαδικασίες, έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερη και πιο δίκαιη κατανομή της δικαιοσύνης. Όπως είπα και πιο πριν, οι ακτιβιστές της Παππούα συλλαμβάνονται και κρατούνται για ειρηνικές διαδικασίες, όπως, ας πούμε, όπως σας είπα η έπαρση της σημαίας ή η συμμετοχή σε δημόσιες ε, δραστηριότητες, όπως το Κογκρέσο των, ε, λαών, των πολιτών της Παππούα. Ε, κατηγορούνται για προδοσία πολλές φορές, σύμφωνα με το 106 του ποινικού κώδικα της Συντονισίας και με σχετικά άλλα τέτοια δικήματα και έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές φορές και φυλάκιση 20 ετών. Σύμφωνα με δεδομένα από τη δική μου οργάνωση υπάρχουν περίπου 30 πολίτες από την Παπούα που, περιμέ... που κρατούνται και περιμένουν να δικαστούν ή ε, είναι ήδη φυλακισμένοι για προδοσία. Πολλοί έχουν ε, φυλακιστεί ήδη από το 2008 και αυτοί που τους φυλάκισαν έχουν ε, να αντιμετωπίσουν ποινές 8 μηνών έως 6 ετών. Ο επικεφαλής ε, του ε, Συμβουλίου της ε, Παπούα που κατηγορήθηκε για προδοσία κατηγορήθηκε ο ίδιος για προδοσία μετά τη συμμετοχή του στο Κογκρέσο των Πολιτών της Παπούα. Ένας από τους, από τους, από τους κρατούμενους είναι επίσης κατηγορείται για προδοσία και καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης ο ΙΕ βρήκε ότι η καταδίκη αυτή παραβιάζει την, ε, τα πρότυπα διεθνών, ε, ε, α, των διεθνών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. και ζήτησε από την Ινδονησία να αποφυλακιστεί, καθώς επίσης και να αποφυλακιστούν όλοι οι υπόλοιποι που κρατούνται παράνομα. Η ελεύθερη τη έκφραση επίσης είναι πολύ σημαντική για, την, για τους πολίτες της Παπούα και για την προστασία όλων των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Επίσης είναι σημαντική ε, απέτηση για την επίλυση των ε, δαφικών προβλημάτων που υπάρχουν. Η επίλυση του προβλήματος αυτού είναι σαφής η κυβέρνηση της Ινδονησίας θα πρέπει να σταματήσει αυτή την πρακτική των, της κατηγορίας με ποινικά, δικαιώ, με δικήματα όπως η προδοσία για, σε άτομα που απλώς συμμετέχουν σε ε, ειρηνικές δραστηριότητε. Πρέπει να υπάρξει ε, ε, ε επίτευξη εμπιστοσύνης για, για μια τέτοια διαδικασία θα ενθάρρυνα αυτή την υποεπιτροπή να μελετήσει με όποιο τρόπο μπορεί και να ασχοληθεί με τα θέματα αυτά, ειδικά σε σχέση και με τον μηχανισμό που υπάρχει για, στα πλαίσια του διαλόγου Ευρωπαϊκής Ένωσης Συντονισίας, ο οποίο γίνεται και στις Βρυξέλλες και στην Τζακάρτα. Επίσης θα ήθελα τα μέλη τη Επιτροπή σα να ελέγξουν τα, το, τι συνέβη, ε, το τι θα συμβεί μάλλον ε, τα, στις, ε, στην επέτειο της 1ης Δεκεμβρίου και να μπορέσουν να, και να παρέμβουν για να αποφύγουμε παρόμοιες κατα, καταστάσεις επιτόπου. Σας ευχαριστώ και πάλι που μου δώσατε τη δυνατότητα να απευθυνθώ σε εσά και βεβαίως ευχαριστώ να σας απαντήσω και σε ερωτήσεις. <clears throat> który niestety odwołał swój przyjazd na dzisiejsze posiedzenie podkomisji praw człowieka ze względu na... να mm, Ο κύριος Νέλε ακύρωσε την παρουσία του εδώ. Η κατάσταση στην ε, Παππού επιδεινώνεται και έχουμε λάβει μία επιστολή. κύριος Μπάρμπερ πρόκειται να κάνει την εισήγηση. This is για αυτό το μήνυμα από τον πατέρα Ταμπέ. Πρώτα-πρώτα θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη διότι δεν μπόρεσα να παραστώ στην συνάντησή σας ε, που είναι τόσο σημαντική. Έλαβα την απόφαση να μην έρθω στις Βρυξέλλες διότι οι αντιπαραθέσεις ε, έχουν ενταθεί στην Δυτική Παπούα και οι κάτοικοι της χώρας τώρα ε, γιατί προετοιμάζουν τον εορτασμό τη 1 η Δεκεμβρίου. περισσοτερε δυναμει ασφαλεια όμω αναπτύσσονται στη Δυτική Παππούα και όλο ένα και περισσότεροι ε, ανησυχούν. Αυξάνεται η αναταραχή και οπότε γι' αυτό διάλεξα να μείνω ε, κοντά στο λαό μου αυτή την κρίσιμη ώρα. Θα ήθελα επίση να σα ευχαριστήσω διότι μου επιτρέψατε να σα πω πώ έχουν τα πράγματα, πώς έχουν οι σχέσει μεταξύ Ινδονησία και Δυτική Παππούα. Η σχέση μεταξύ τη κυβέρνηση, τη Τζακάρντα και το κατοίκων τη Παππούα ε, ήταν και είναι ακόμα σχέση ε, αμοιβαίας ε, υποψίας, καχυποψίας και δυσπιστίας. Η Δυτική Παππούα, σύμφωνα με αυτή την κατοχή τώρα, έχει γίνει μια χώρα βίων αντιπαραθέσεων και αυτό πηγάζει από, την, από τις διαφορές όσον αφορά την προσάρτηση της χώρας στην Δημοκρατία της Ινδονησίας, που θεωρεί ότι είναι τμήμα της επικρατείας της Δυτική Παππούα και θεωρεί ότι είναι και πρέπει να παραμείνει επομένως κομμάτι της επικρατείας της χώρας και γι' αυτό η αντίσταση θεωρείται απειλή εις την εδαφική ακυρότητα της Ινδονησίας. Η εκρίζωση αυτού του αποσχιστικού κινήματος στη Δυτική Παππούα ήταν ε, ο λόγος που προκάλεσε την κρατική βία και καταστολή κατά των κατοίκων της ε, Παππούα, των παραδιάσεων των δικαιωμάτων που έχουν γίνει κατά των Ιθαγενών και γι' αυτό νομίζω ότι μάλλον θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και στο μέλλον, διότι χιλιάδες στρατευμάτων έχουν αποτυχθεί στη χώρα και η αιτία του προβλήματος δεν έχει φυγεί, δεν έχει αντιμετωπιστεί. Στο μεταξύ, πάρα πολλοί από τους ε, κατοίκους της χώρας βλέπουν ότι η χώρα των προγόνων τους ε, τελεί υποκατοχή, κατοχή Ινδονησιακή και θεωρούν ότι είναι απικία της Δημοκρατίας Ινδονησίας και για αυτό και ε, έχουν οργανώσει αντίσταση κατά της επικοινωνικής δύναμης. Αυτή η, η αντίσταση ασκείται με μέσα βία αλλά και ειρηνικά και θα συνεχιστεί επομένως αυτή η αντίσταση του κατοίκων της Παππού. Νομίζω ότι ήρθε τώρα η ώρα η κυβέρνηση να προβληματιστεί και να σταματήσουν παραβιάσεις των δικαιωμάτων και θεωρώ ότι θα ε, γίνουν ακόμα περισσότερες παραβιάσεις των δικαιωμάτων εάν δεν ε, αντιμετωπιστεί η ρίζα του κακού, η αιτία για την οποία έχουμε αυτό το αποσχεστικό κίνημα στη χώρα και αυτό θα πρέπει και δύο πλευρέ με επικοδομητικό διάλογο να δουν ε, τις πραγματικές για του προβλήματο και χωρί ε, περισσότερη αιματοχυσία να προχωρήσουν σε επίλυση. Τα καλά νέα είναι ότι υπό την αιγίδα του Προέδρου του Σύλλογου Μπαμάκλου και οι κάτοικοι τη Παππούα έχουν πει ότι προτίθενται να κάτσουν στο βέστη του διαλόγου για να βρεθεί μια ειρηνική λύση. Ο πρώτος Γιούντο Γιώνο έχει δεσμευτεί ότι μέσω διαλόγου θέλει να λύσει το πρόβλημα και ανεκκίνωσε ότι δεσμεύεται η κυβέρνησή του να κάνει να διαπραγματεύσεων και να ζητηθούν κάποιε λύσει και τα προβλήματα να τείνουν να επιληθούν. Και γι' αυτό και παρακαλώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία για να ανοιχτό διάλογο με του κατοίκου τη Παπούα, ούτω ώστε ειρηνικά να διευθετηθεί το πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί επίση να βοηθήσει, μπορεί να παράσχει αρρωγή, ούτω ώστε η κυβέρνηση στην Ινδονησία να καθίσει για να διαπραγματευτεί, να συνοηθεί με του κατοίκου τη Παππού με ένα ανοιχτό διάλογο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κατανόησή σα και την προσοχή σας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Και ευχαριστούμε που μας αναπτύξατε τόσο έχει να πει ο πατήρ Τιμπέη. Γιατί στην επιστολή του το μήνυμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο για τόσα λέει εδώ πέρα για την επίλυση του προβλήματος. Οπότε μπορούμε παρά να ευχαριστήσουμε τον ε, ιερέα και δεν μπορούμε παρά να του προσφέρουμε την αμέριστη υποστήριξη μας. Και τώρα θα δώσουμε τώρα το λόγο στην κυρία Κόρμπερ η οποία έχει συνεργαστεί με τον κυβερνήτη Τατζέ και έχει συγγράψει με διδακτορική μελέτη όσον αφορά την κατάσταση στη Δυτική παπουά. Είναι εμπειρογνώμων, Είναι ειδική όσον αφορά τα θέματα αυτά. Είχαμε κάνει μια αποστολή 2005-2006 επιτόπου και η αποστολή εκείνη είχε σκοπό να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του Ελσίνκη εκεί. Και η κυρία Κόρμπερ από τότε είχε ασχοληθεί με το θέμα και τώρα θα μας περιγράψει το πώς έχει η κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ έχει αναπτύξει σημαντικό ρόλο, έχει βοηθήσει σημαντικά στη συνεργασία με την κυβέρνηση της χώρας Κόρμπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και αγαπητά μέλη της Υποπιτροπής που μου δίνετε ευκαιρία να σας αναπτύξω το θέμα ε, που αφορά τη Δυτική Παπούα. Σε αδρές γραμμές θα σας αναπτύξω τα εξής. Πρώτα-πρώτα θα προβώ σε κάποια σύνοψη για τα συμπεράσματα που έχουμε αντιλήσει από τη διαδικασία που κράτησε 6 διαδικασία ΑΤΣΕ και κατόπιν θα δούμε ποιε είναι οι επιπτώσεις για τη χώρα κατόπιν αυτών δηλαδή των ε, διαδημάτων. και ε, επίσης θα σας πω για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να κάνει κάτι ε, συνεργαζομένη με κάποιον διαμεσολαβητή από έξω. Ξεκίνησαμε λοιπόν αυτό το, το μνημόνιο που αφορούσε την, το, την κυβέρνηση της χώρας και, την, την, και το κίνημα Ατσέχ. Αυτό έγινε τον Αύγουστο του 2005 και αυτό θεωρήθηκε τότε ότι αποτελεί μια επιτυχία. Αυτό επίσης ε, ισχύει το στο μάλλον διότι από τότε έπαυσαν οι παρεμβάσεις των δικαιωμάτων. Παρ' όλα αυτά όμως αυτή η διαδικασία της ειρήνευσης δεν οδήγησε σε απόδοση ευθυνών για τις ε, παρελθούσες παραβιάσεις των δικαιωμάτων. Ούτε επελήφθη η Επιτροπή των Δικαιωμάτων, ούτε η Επιτροπή για την Αλήθεια και τη Συμφιλίωση. Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς να πει ότι έμαθε τίποτα αν τις κάποια χρήσιμα συμπεράσματα από αυτή τη διαδικασία τσεκ όσον αφορά την απόδοση ευθυνών για την παραβίαση αυτών. Τώρα, τους ε, πρώτους 15 μήνες η υλοποίηση αυτού του μνημονίου του Ελσίνκη παρακολουθήθηκε από την ε, σχετική Επιτροπή Εποπτείας και Παρακολούθησης ε, όπου συμμετέσχουν και πέντε χώρες του ΑΣΕΑΝ. Συμφώνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει μια ειρηνευτική αποστολή και ότι δεν ήθελε να εμπλακεί ο ΟΗΕ διότι, διότι θεωρεί το μεροληπτική συμμετοχή του ΟΗΕ εις ε, την υπόθεση της ε, εξαρτησία του Ανατολικού Τιμόρ και έχουμε ότι αυτές την πρώτη, ε, τον πρώτο αφοπλισμό ε, της, της ΓΑΜ και οπότε και τα δύο μέρη που είχαν προσφοράσει το μνημόνιο του Ελσίνκη επιβεβαίωσαν ότι αυτή η αποστολή που και παρακολούθησης επιτυχώς είχε εκτελέσει την εντολή της. σε σχέση με την εντολή του είχε δώσει ο ΙΕ δηλαδή, και ακόμα έπρεπε να συμμορφωθεί με το μνημόνιο η κυβέρνηση της χώρας. Έχουν περάσει πέντε χρόνια και αυτά ακόμα δεν έχουν γίνει. Εγώ έχω, ε, διδάχθηκα τα εξή, δεν τα εξής συμπεράσματα από τη διαδικασία ειρήνευση τη ΑΤΣΕΧ. Ότι η πολιτική βούληση για να περτανεύσει ειρήνη ήταν ε, δεδομένη. Και ο τότε αντιπρόεδρος Γιουσούφ Κάλα ε, λιγανά είχε δεσμευτεί. Κατά το εξάμεινο των ειρηνευτικών ε, διαδικασιών και συνομιλιών ανέλαβε τις ευθύνες ο Κάλα ούτως ώστε να, να καλύψει τα αιτήματα της, ε, του, της ΓΑΜ, της, ε, της, του, του, του κινήματος και πέρασε το 2006 ένας, μια, μια ειδική νομοθεσία ε, που προέβλεπε εκτεταμένη αυτονομία και επίσης κατά δεύτερο λόγο ε, και το κίνημα ΓΑΜ ε, συνοήθηκε με τον, με τον κυβερνήτη Ιρβάντι Ιουσούφ και παρόλα αυτά όμως η ηγεσία του κινήματος έμεινε στο εξωτερικό και προσπάθησε να παρεμποδίσει την ομαλή πρόοδο της εφαρμογής του μνημονίου. Είχαμε πάρα πολλές δωρεές που έφτασαν μετά το χτύπημα από το τσουνάμι σε πάρα πολλά δις αμερικανικά δολάρια για την ανασυγκρότηση της χώρας. Και επομένως ανέλαβε το κίνημα να ανασυγκροτήσει τη χώρα περισσότερο από ότι η κυβέρνηση που δεν λειτουργούσε. Στο δε Ελσίνκι η αποστολή εποπτεία, μάλλον το κίνημα, το κίνημα Τσέχ, θεώρησε ότι μπορεί να κατέβει στις εκλογές όταν γίνουν. Από το 2007 και 2009, ε, αφού κέρδισε τις εκλογές, βρίσκεται στην κυβέρνηση και καθορίζει τον πολιτικό βίο της χώρας και σε εκτελεστικό και σε νομοθετικό επίπεδο. Υπάρχουν ε, κάποιοι πόροι που ζουν στη χώρα, φτάνουν ε, το 1 δις δολάρια ετησίως. Οπότε πια οι ντόπιοι πολιτικοί δεν μπορούν να κατηγορούν την Τζακάρτα όπως το παρελθόν ότι ευθύνεται για την υπανάπτυξη της ε, χώρας. Η δε ε, αποστολή εποπτείας αντιστάθμιζε τις αδυναμίες των ε, δύο αντιπάλων μερών και έγινε, έγινε προσπάθεια να κάτσουν τα αντίπαλα μέσα των διαπραγματεύσεων τώρα. Όσον αφορά τις συνέπειες για τη Δυτική Παππού, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι το κίνημα ειρήνης δεν ταυτίζεται με τη χώρα και ότι το μοντέλο της ειρήνευσης δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί 100%. Αν το κάνει κανείς αυτό θα είναι αντιπαραγωγικό. Θα πρέπει να, επισημάνουμε τις διαφορές της Δυτικής Παππούα από ΑΤΣΕ και να αναγνωριστούν οι ιδιομορφίες της Δυτικής Παππούα να δούμε το ιστορικό πλαίσιο ότι ανέκαθεν υπήρχε ε, δυσπιστία προς την ε, δημοκρατία της Ινδονησίας. Μιλούμε για 240 εθνότητες που συναπαρτίζουν τη χώρα, οπότε γι' αυτό και είναι άκρος ετερογενής ε, και οπότε γι' αυτό και έχουμε και ένα σωρό εσωτερικές προστριβές. οι κάτοικοι της Παππούα είναι ως επιτοπλίστων χριστιανοί και θεωρούν ότι έχουν περιθωριοποιηθεί από την μαζική εισρωή ε, εξωτερικών στοιχείων που οι περισσότεροι είναι Ινδονήσοι και Μουσουλμάνοι. Οπότε το θέμα τώρα έχει και θρησκευτική πτυχή και πολλοί από τους κατοίκους της Παππούα φοβούνται ότι προβαίνει σαν στρατηγική ελέγχου, σαν καπέλωμα ε, τον εξισλαμισμό η κυβέρνηση της Τζακάρτα. Κάτι, και αυτό το σχετικό στοιχείο άκουσε στο παρελθόν. Ε, τώρα έχουμε όλες αυτές τις εσωτερικές ε, προστριβές που είναι πάρα πολύ πολύπλοκες. Και αυτό επηρεάζει τις σχέσεις και με την Τζακάρτα και με το κίνημα της αντίστασης. Και η κατάσταση τώρα είναι πολύ πιο πολύπλοκη από ότι η από ότι το, το πώς ήταν η κατάσταση με το κίνημα μέχρι το 2006. Πάντως, τώρα δεν, βοηθά, δεν βοηθούν οι εκπρόσωποι ε, του κινήματος ε, ΓΑΜ της, την διαδικασία. Πάντως, επίσης, ο νόμος 21 του 2001 για την ειδική αυτονομία ε, μοιάζει πάρα πολύ με τον ειδικό νόμο της αυτονομίας του 2001 και αυτό ε, βέβαια έχει να κάνει και με το πόσες αρμοδιότητες έχει ή δεν έχει εκχωρήσει ακόμα η κυβέρνηση της Τζακάρντα. Όσον αφορά την ΑΤΣΕΧ και το 2001 και το 2006 ε, δεν είχαμε και τίποτα ε, εκτεταμένες παραχωρήσεις αυτονομίας και η διαφορετική ε, και η μεγαλύτερη διαφορά αφορά ε, την εφαρμογή αυτού του νόμου, αυτή, την ε, νομοθεσία του 2006. Δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία με την ε, Τζακάρντα που να μοιάζει με το μνημόνιο του Ελσίνκη. Πάντως, συνεχίζει και υπάρχει ε, δυσαρέσκεια και από το, τις παραχωρήσεις της Τζακάρτα και από το κατά πόσον τηρεί Τζακάρτα συμπεφωνημένα. Η κυβέρνηση της 2006 από τότε που έφυγε η αποστολή παρακολούθηση κάνει τα εξή. Χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιτεύχθηκαν πολλά. Είπαν όμω ότι από εδώ και στο χρειαζόμαστε και θα κανονίζουμε τα, τα, του οίκου μα μόνοι μα. Αυτό τι πάει να πει. Ότι δεν έχει πολιτική βούλη στην Τζακάρτα, ούτω ώστε κάποιο εξωτερικό δημοσιολογητή να παρέμβει στη σχέση με τη Δυτική Παπούα. Και επίση, ε, αυτό το βρίζει μια ιστορική δυσπιστία προς τους ε, ξένους. Είναι πεπισμένοι ότι μπορούν από μόνοι τους να καταφέρουν αυτά τα οποία είχε καταφέρει η, η αποστολή ε, παρακολούθηση σε σχέση με το ΑΤΣΕΧ. Νομίζω ότι αυτό είναι μια υπερεκτίμηση των δρατοτήτων τους. Με τίποτα δεν πρόκειται να καταφέρουν να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι όλοι οι εμπλεκόμενοι ακριβώς όπως είχε καταφέρει να κάνει η αποστολή παρακολούθησης σε 44 συναπτές συναντήσεις. Παρ' όλα αυτά δεν θα πρέπει να χάνουμε χρόνο με τα λόμπι ε, και να δούμε κατά πόσο υπάρχει περιθώριο το Ηνωμένα Έθνη ή διεθνή μη κυβερνητική οργάνωση να διαδραματίσει έναν ρόλο στην Ατσέχο όπως έκανε η αποστολή της εποπτείας και έτσι να δούμε κατά πόσο είναι δυνατόν η κυβερνητική οργάνωση να ασκήσει ένα ειδικό βάρος όπως έκανε κάποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα, τα τη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν πάρα πολύ θετικός καταλήτης για την ειρηνευτική διαδικασία, όμως η εντολή ήταν περιορισμένη και κυρίως αφορούσε την οικονομική και κοινωνικοπολιτική ε, διάσταση του θέματος. Τώρα είναι το διακύβημα πολύ ευρύτερο Χρειάζεται η Τζακάρτα από τώρα και για πολλές δεκαετίες να προσπαθήσει ε, πάρα πολύ σοβαρά. Γι' αυτό νομίζω ότι αν υπάρχουν κάποιο είδους ε, ψύχρεμες ε, συνεννοήσεις μεταξύ Τζακάρτα και Δυτικής Παππούα θα προχωρήσουμε σε κάποια διάσκεψη ειρηνευτική. Ο πρόεδρος χρησιμοποίησε αυτό το μήνα τη λέξη διάλογος και θα πρέπει βέβαια να συγκεκριμενοποιηθούν οι συνοήσεις, αλλά νομίζω ότι έχουμε την απαρχή ενός ε, θετικού πλαισίου. Επίσης νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλό από το μέρους του Προέδρου το ότι απεφυλάκησε κάποιους ε, ε, πολιτικούς κατουμένους οι οποίοι είχαν καλή διαγωγή. Στο ΑΤΣΕΧ υπήρχε ομοφωνία στην Παπούα παρά το ότι υπάρχει αυτή η μονάδα για την επιτάχυνση της ανάπτυξης, εκεί υπάρχει ε, πολυφωνία, εκεί δεν ακούγονται θέτους ε, με μηνύο τρόπο και δυστυχώς φαίνεται ότι η κυβέρνηση της Ινδονησίας δεν διδάχτηκε τίποτα από την θετική εμπειρία της ειρηνευτικής διαδικασίας. σταμάτησε τώρα η καταστολή όπως το και αστυνομία. όμω, από ό,τι μαθαίνουμε, οι δυνάμει ασφαλεία, εκεί ε, είναι μισθέ από τον κόσμο. Άρα, με αυτόν τον τρόπο δεν γίνεται τίποτα. Εκτός εάν αποχωρήσουν ακόμη περισσότερο. αυτά που κάποτε έκανε η Δονησιακή αστυνομία, τώρα τα κάνουν αυτές οι δυνάμεις που βρίσκονται στη χώρα και επομένω δεν έχει σημειωθεί και πολύ μεγάλη πρόοδος. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κόρμπερ, για όλα αυτά τα τόσο ενδιαφέροντα τα οποία μας εξηγήσατε. για παπούα και για Ατσέχ. Μας τονίσετε ποιες είναι οι διαφορές ε, στις δύο καταστάσεις. Και τώρα έχουμε τον κύριο Βάργας που εκπροσωπεί την εξωτερική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει ανάψει το μικρόφωνο. Is that okay now? Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, που προσκαλέσατε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να παρευρεθεί στη συνάντηση αυτή. Και θέλω κάπως σύντομα να σας μεταφέρω κάποιες σκέψεις της υπηρεσίας μας για την κατάσταση στην Παπούα και κυρίως όσον αφορά τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ινδονησία. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης παρακολουθεί όσο μπορεί πιο στενά την κατάσταση στις επαρχίες της Παπούα και της Δυτικής Παπούα με επαφές, με μη κυβερνητικέ οργανώσεις, με άλλους παράγοντες αλλά και μέσω των αποστολών που έχει με ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες, δηλαδή στην Τζακάρτα. Τα τελευταία βία γεγονότα που έλαβαν χώρα τον Οκτώβριο που μας πέρασε και που κατέληξαν σε θανάτους μεταξύ του πληθυσμού είναι θέματα που προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο αυτή έχει θέσει στον ε, αρμόδιο υπουργό στη Τζακάρτα και στις διάφορες επίσημες συναντήσεις που έχουν λάβει χώρα στην Ινδονησία τον Νοέμβριο, 14 Νοεμβρίου. Μάλιστα με την ευκαιρία αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράμμισε την αναγκαιότητα να γίνουν αμερόληπτες έρευνες για, ε, για τους θανάτους ε, αυτούς που προκλήθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Θέλω εδώ να ξεκαθαρίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται την εδαφική ακαιρεότητα της ε, Ινδονησίας μέσα στα σημερινά της σύνορα και δεν στηρίζει αποσχιστικά κινήματα στην Παππούα. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί για τις εξελίξεις στην Παπουά, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν τηρούνται όπως για παράδειγμα η ελευθερία έκφρασης, η ελευθερία του συναθρίζεστε ειρηνικά, αλλά επίσης επειδή υπάρχει υπερβολική χρήση βίας από πλευράς των αρχών εκεί. Αδιαφυσβήτητα, όπως το είπαν και άλλοι ομιλητές εδώ, η Ινδονησία έχει βελτιώσει την ε, προστασία της και το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Παραμένουν όμως θέματα για ανησυχία. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ιδανησία χρησιμοποιεί το μέσο που διαθέτει για πολιτικό διάλογο ώστε στα πλαίσια αυτά να θέτει τα ζητήματα που μας απασχολούν και πιέζουμε την κυβέρνηση να φροντίσει για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την τιμωρία των υπευθύνων που τα παραβιάζουν. Τώρα εδώ στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε το θέμα του βασανισμού φυλακισμένων από την Παπούα. Ο κ. Μπάρμπερ αναφέρθηκε σε αυτό. Όπως επίσης και για τις ποινές οι οποίες επιβάλλονται ε, από στρατιωτικά δικαστήρια για προδοσία κλπ. Εμείς ενθαρρύνουμε την κυβέρνηση της Δονησίας ε, να συνεργαστεί με τον πληθυσμό τους αυτόχθονες της Παπούα όσον αφορά τον νόμο αυτονομίας και την εφαρμογή του νόμου του 2001 για αυτονομία της Παπούα. Φυσικά και θέλουμε να υπάρχει καλή διαχείριση των θεμάτων αυτών στην ε, Παπούα. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστηρίξει και τα τελευταία βήματα τα οποία έχει κάνει η κυβέρνηση της Ινδονησίας με εκπροσώπους από την Παππούα όσον ε, αφορά την εμπλοκή των αυτοκτόνων στις πολιτικές εξελίξεις με συμμετοχή και εκπροσώπων των ε, Υπουργείων. Μια τέτοια συνάντηση έγινε τον Ιούλιο που μας πέρασε για παράδειγμα. Εμείς βλέπουμε να υπάρχουν θετικές εξελίξεις στη Τζακάρτα με την τελευταία δήλωση του Προέδρου Χογιώνο, ο οποίος είπε ότι η κεντρική κυβέρνηση είναι ανοιχτή στο διάλογο. Χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό, γι' αυτήν την ε, διάθεση τη θετική που εκφράστηκε και που ενθαρρύνεται και από τη δημιουργία μιας νέας ε, ομάδας στην οποία θα συμμετέχουν αξιωματούχοι στην Χαραπούτα και στο Κανιμάρι. Επίσης λαμβανόμαστε ότι αυτή η νέα μονάδα θα συντονίσει τις νέες προσπάθειες που γίνονται στην Ινδονησία, αλλά θα ασχοληθεί και με τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα δουλέψει η μονάδα αυτή. Τώρα ίσως σας ενδιαφέρει να μάθετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί διάφορα προγράμματα ανάπτυξης στην ε, Παππού και τη Δυτική Παππούα όσον αφορά την εκπαίδευση για παράδειγμα για να μειωθούν οι μεγάλες διαφορές που υπάρχουν στα επίπεδα ε, εκπαίδευσης στην περιοχή. Όπως επίσης δουλεύουμε και για να αντιμετωπίσουμε διαφορές μολυσματικές ασθένειες. Συχνά πρόκειται για μικρά προγράμματα τα οποία έχουν ως στόχο να στηρίξουν την κοινωνία των πολιτών υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προκειμένου σιγά σιγά να περάσουμε σε ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα για τις κλιματικές αλλαγές στην Παπούα. Για να συνοψίσω λοιπόν, θα ήθελα να επαναλάβω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τον επικοδομητικό διάλογο ανάμεσα στους εκπροσώπους της Παππούα και την κυβέρνηση της Ινδονησίας προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδο και σε επίπεδο της νέας μονάδας που δημιουργείται. Αλλά τονίζω συγχρόνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να ζητάει πρόσβαση στις επαρχίες Παππούα για τους ε, διπλωμάτες, για αμερόληπτες ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, όπως για παράδειγμα για την ε, Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού. Αλλιώς ε, δεν πιστεύω ότι εξυπηρετούνται ούτε τα συμφέροντα της Ινδονησίας. Συνεχίζουμε επίσης να θαρρύνουμε την κυβέρνηση της Ινδονησίας προκειμένου να προβεί σε αμερόληπτες έρευνες σχετικά με τις δολοφονίες που έλαβαν χώρα από τις υπηρεσίε ασφαλείας και για την τιμωρία των υπευθύνων. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Βάργα. Σας ευχαριστούμε που παρουσιάσατε την άποψή σας. Η κυρία Γελμπός θέλει να παρέμβει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να παρέμβω. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές που θα μας, μας έδειξαν έτσι ένα, μια, μας έδωσαν μια μερική εικόνα της κατάστασης των προβλημάτων. Νομίζω ότι ένα μέλος εδώ του Κοινοβουλίου όπως εγώ που ε, δεν έχω ασχοληθεί με το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη περιοχή του κόσμου, περισσότερο με άλλα μέρη της Ασίας, αλλά ε, σήμερα δεν έχω έτσι, μια γενική ε, εικόνα της κατάστασης. Απ' την άλλη, ως Γερμανίδα βουλευτής, Είμαι πάντα σε επαφή με τις εκκλησίες μας, με οργανώσεις στον τρίτο κόσμο κτλ. Και λαμβάνουμε κάποιες πληροφορίες που μας κάνουν να σκεφτούμε. Ποια είναι τα ερωτήματα που θα μπορούσαμε να σας θέσουμε. Ειδικά σε ό,τι αφορά το ERT. Συγκεκριμένο ερώτημα λοιπόν. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε παραπάνω για, την, ε, για μια διαδικασία συμφιλίωσης. Μιλήσαμε για προβλήματα συνύπαρξης, για προβλήματα σε όλη την αναπτυξιακή διαδικασία, ε, σε μια έτσι, παράθεση των γεγονότων για το τι μπορεί κανείς να παρατηρήσει κτλ και τι μπορεί να κάνει ή να μην κάνει. Αλλά εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, η ευρωπαϊκή οικονομία ποια είναι, τι θέση έχει απέναντι σε αυτή τη χώρα. Και με βάση αυτό δεν μπορούμε να δούμε μόνο τις οικονομικές πτυχές και δεν ξέρω αν το κάνουμε ε, ούτως ή άλλως αυτό ένα κομμάτι της ερώτησής μου είναι αυτό, αλλά εμείς ως ε, Ευρωπαίοι βουλευτές έχουμε την ε, υποχρέωση να, να δούμε τι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είπατε τις τελευταίες εβδομάδες ε, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν. Μου είπαν και οι εκπρόσωποι μας εκεί και εκπρόσωποι εκκλησιών κλπ. ότι ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί πολύ εν τω μεταξύ. Και βεβαίω θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τον σεβασμό προ του αυτόχθονες, οι οποίοι είναι χριστιανοί κατά το πλήστον. Εμείς πώς μπορούμε, τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω. έτσι ώστε αυτό το πρόβλημα να μπορέσουμε να το επηρεάσουμε θετικά, να δώσουμε μια προοπτική στους ανθρώπους. Και βεβαίως όχι απλώς να πούμε στους υπευθύνου της χώρας ε, είναι λάθος αυτό που κάνετε, αλλά να βρούμε ένα, ένα τρόπο να λύσουμε το πρόβλημα. Αν, εδώ, ε, αν είχαμε την Αραβική Άνοιξη ε, σε τέτοιες κοινωνίες που είδαμε να συμβαίνει, νομίζω ότι θα μπορέσουμε και εδώ να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός. Γιατί η κατάσταση εκεί φαίνεται ότι δεν είναι εύκολη, μάλλον είναι αρκετά περίπλοκη. Νομίζω όμως ότι πρέπει να αναρωτηθούμε ποιες είναι οι συνέπειες, οι συγκεκριμένες συνέπειες ε, αυτών των ε, διαμαχών και σε ό,τι αφορά την κοινωνική πτυχή, για τους ανθρώπους δηλαδή, και για την οικονομική πτυχή, αλλά και για τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, επιτόπου. Ποια είναι η κατάσταση αν μου πείτε ότι 40 άτομα, 40 χριστιανοί έχουν σκοτωθεί την, ε, τις προηγούμενες εβδομάδες, ε, προφανώς αυτό το πράγμα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Έχω την εντύπωση ότι θέλατε να μας πείτε ότι έχουμε λίγες πιθανότητες ή λίγες δυνατότητες να δράσουμε. Αυτό είναι, το, ε, αυτό είναι αυτή είναι η πραγματική κατάσταση. Ευχαριστώ. E, Ευχαριστώ. Να δώσουμε πάλι τον ε, λόγο στην EAD. Και θα δώσουμε και τον ε, λόγο στον ε, πρεσβευτή της συντονισίας. Νομίζω ότι το θέμα είναι η πρόσβαση και για μη κυβερνητικές οργανώσεις και για άλλους. Πώς δηλαδή μπορούμε να διευκολύνουμε επιτόπου την κατάσταση. Πρέπει και εμείς να δούμε πώς έχει η κατάσταση με τα μάτια μας. Και γι' αυτό πρέπει να δούμε ποια εμπόδια τελικά υπάρχουν που δεν μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Το είπε βεβαίω και ο πρόεδρος της Ινδονησίας ότι θα πρέπει να επιστρέψουμε στα πλαίσια του διαλόγου. Αλλά αυτό γιατί δεν είναι δυνατόν στην Δυτική Παππούα, γιατί δεν γίνεται να βρεθεί μια, μια ειρηνική λύση. Προφανώς υπάρχουν ε, διαφορές, μας τα είπε και η κυρία Μπάρμπερ. Υπάρχουν διαφορές ό,τι αφορά τη θρησκεία. Ε, εντάξει, αυτά, αυτό προφανώς είναι σημαντική διαφορά ε, και σημαντικός παράγοντας που προφανώς ε, τροφοδοτεί τα, τις διαμάχες. Μιλούμε και για την τιμωρία όσων όντως πρέπει να τιμωρηθούν. Και εδώ θα μπορούσα και εγώ να σας πω για την ε, δική μου εμπειρία. Ε, προφανώς ε, το να αντιμετωπίσουμε το παρελθόν παίζει σημαντικό ρόλο για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και το παρόν. Βεβαίω υπάρχουν ακόμη και, σήμερα στην Πολωνία δικαστικέ διαδικασίε που εκκρεμούν από τον ε, ε, καιρό της, ε, του κομμουνισμού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να γίνει ένα πρώτο βήμα. Για να μπορέσουμε τελικά να συνεννοηθούμε όλοι μεταξύ μας. Πρέπει να υπάρξουν, υπάρχουν μάλλον πολλές προσπάθειες για ανεξαρτησία. Πρέπει όμως να δούμε πώς όλα αυτά μπορούν να συγκεραστούν. Βεβαίως ε, η Ινδονησία έχει εδώ να παίξει σημαντικό ρόλο. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα βήμα που πρέπει να δώσουμε ε, προς την ε, προς τον πληθυσμό της Παππούα. Το, το πρόβλημα προφανώς είναι πολυσχηδές, είναι επίκαιρο και γι' αυτό τίθεται και το ερώτημα των προσφύγων. Πολλές χιλιάδες προσφύγων που περνούν στην Ινδονησία και διαμένουν εκεί παράνομα και δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν γιατί χρειάζονται οικονομικοί πόροι για να δοθεί το... για να νομιμοποιηθεί ένας πρόσφυγας που ζει στην Ινδονησία. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι ζουν πραγματικά σε μια φαία ζώνη. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Δίνω λοιπόν τώρα το λόγο το... στον κύριο Βάργας. Um, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τα ερωτήματα έχουν τεθεί απαιτούν μακροσκελής απαντήσεις. Πάντως, θα βοηθούσε εάν τονίζαμε κάποιες πτυχές που θα φώτιζαν αυτό το περίπλοκο θέμα της Δυτικής παππού που είναι μια πραγματικά δύσκολη περίπτωση. Και πάλι σας τονίζω το εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτα-πρώτα θέλει να αντιμετωπίσει τα θέματα τα σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ο διάλογος, ο οποίος ξεκίνησε εδώ και κάποια χρόνια, είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό για αυτή την υπόθεση, γιατί νομίζω ότι έτσι μπορούν και οι μεν και οι δε να θέσουν επί τις τραπέζες με τρόπο ειλικρινή τα θέματα τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν. Και εγώ σας τονίζω πόσο χρήσιμη υπόθεση είναι αυτός ο διάλογος. Ιδίως για τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και στην Παππού και στη Δυτική Παππού. Υπάρχει το θέμα βέβαια της ε, χρηστής και το οποίο προσπαθούμε να το διεκπαιρεώσουμε. Πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με κάποια προγράμματα συνεργασία που έχουμε με τη χώρα και αφορούν την Παππούα και τη Δυτική Παππούα. Όπω προείπα, εμεί είμαστε αναφαντών υπέρ του διαλόγου. Και όσον αφορά το ότι θα πρέπει να δεσμευτεί η κεντρική κυβέρνηση της ε, Τζακάρτα ότι θα συνεχίσει με συνέπεια τις συνομιλίες με τους εκπροσώπους του λαού της Παπούα. Θα πρέπει να σταματήσει η αμοιβαία δυσπιστία και πάλι τονίζουμε επομένω πόσο σημαντικός είναι ο διάλογος και πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθάει. Δεν θα πρέπει κανείς πάντως να παραβλέπει ότι αυτό είναι θέμα εσωτερικό μην παρεξηγείτε όμως αυτό, διότι η διεθνής κοινότητα κάνει ό,τι μπορεί, ούτως ώστε να βοηθά το να υπάρχει η ευθυντική κυβέρνηση στη χώρα. Οπότε και εμείς θεωρούμε ότι βρίσκουν ανταπόκριση αυτά τα οποία πρόθυμα. έχουμε ε, προχωρήσει όσον αφορά τις επαφές, το διάλογο, ούτω ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορούμε να σταματήσουμε δυσμενείς διακρίσεις με τη βάση θρησκείας που ήταν κάτι το οποίο είχε απασχολήσει πάρα πολύ. Έχει τεθεί και συζητηθεί το θέμα μέσω του προαναφερθέντος διαλόγου. με κάθε ευκαιρία. Και εδώ θα βάλω τελεία. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μαρτίνες Βάργας. Τώρα, κύριε Πρέσβη, έχετε εσείς τη σκητάλη. Εξοχότατε για να προσοφιάσετε τις απόψεις σας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να απευθυνθώ στα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής σας. Μου είναι δύσκολο τώρα να θίξω ένα τόσο περίπλοκο θέμα με μια τηλεγραφική παρέμβαση, αλλά να σας πω κάποια βασικά σημεία που η χώρα μας θα ήθελα να σας εκθέσει. Τότε που σταμάτησε η απεικιοκρατία ε, με, με δυσκολία γιατί δεν ήθελαν με τίποτα να φύγουν οι Ολλανδοί ε, από τότε έχει ενδιαφέρον η αρχή διεθνούς δικαίου που λέει ότι, ότι τα νέα ε, κράτη τα οποία ανεξαρτοποιούνται μετά την αποχώρηση του, του απεικιοκράτη κληρονομούν την επικράτεια που είχε ο απεικιοκράτης. Η δύναμη τέλο πάντων. Και εν προκειμένου αυτό έσχισε όσον αφορά την Ολλανδική επικοκρατία. Οπότε και εμείς δεν βλέπουμε πώς ε, ε, ε κατόπιν της δυσκολίας των που είχαμε για να αποχωρήσουν. Οπότε, και σε σχέση με την Αφρική. Επιβεβαιώθηκε αυτή η αρχή του διεθνού δικαίου ότι δηλαδή τα βιοκρατικά σύνορα γίνονται τα σύνορα του νέου εξάρτητου κράτου. Επομένω, όπω είπε πολύ καλά την ιστορία μα, είχαμε ε, ε, καταστολή, είχαμε πάρα πολύ αυταρχικό κράτο από τη δεκαετία του 60, έλεγχος των ΜΜΕ, ε, καταστολή κάθε ελευθερίας. Γι' αυτό και δεν θεωρούμε ότι με αυταρχικό τρόπο είναι δυνατόν να επιληθεί κανένα θέμα, ούτε το θέμα της ε, Παππού. Υπήρχε ένας ειδικό νόμος του 2001. Αυτός προέβλεπε ειδική αυτονομία για την Παπούα. Να σας πω τα βασικά στοιχεία αυτού του νομοθετήματος. Πρώτα-πρώτα ότι η περιφερειακή κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή, έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την διακυβέρνηση της χώρας, εκτός από την εξωτερική πολιτική, την αμυντική πολιτική και την εθνική άμυνα και κυβέρνητες και, αντι, και, και μπορεί να είναι μόνο κάποιος που προέρχεται από τη χώρα. Έγιναν οι εκλογές και είχαμε τέσσερις υποψηφίου. ε, 600.000 ψήφισαν σε 2.000 εκλογικά κέντρα και ήταν τέσσερις υποψήφοι που είπαν τοπική. Οπότε εξελέγει αυτή η τοπική κυβέρνηση και τοπική βουλή στην Ινδονησία δεν προβλέπεται άλλο τέτοια τοπική περιφερειακή κυβέρνηση ε, και έχουμε κάποια άρθρα σε αυτό τον νόμο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίση συγκροτήθηκε αυτή η Επιτροπή για την ε, Συμφιλίωση και αυτό προτάσει τη κυβέρνηση. Ο της οικονομική, τώρα κύριε Πρόεδρε, δυνάμει αυτού του δικαίου η Παπούα ε, ελέγχει 80% από τα εισοδήματα από γεωργία, δάση, αλεία. 70% από φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Είναι η μόνη επαρχία στην Ινδονησία που έχει τέτοια δικαιώματα. Η άλλη είναι η Άτσε. Οι άλλες επαρχίες έχουν μόνο 15% του, του, των εσόδων από φυσικό αέριο και πετρέλαιο. 90% επίσης των φόρων των σχετικών με την πράγματι ε, παραμένουν στον κορβανά της χώρας το εισόδημα της χώρας ήταν 5-3 ε, τοπικού νομίσματος. Το 2010 έγιναν 10-3. Το 2008 15-3 δηλαδή 6,1 δις δολάρια. Ο πληθυσμός είναι 4 εκατομμύρια σχεδόν. Αυτό σημαίνει ότι το ΑΕΠ της Παππούα το 2008 ήταν σχεδόν 7.000 δολάρια 10 φορές πιο πολύ από το Ανατολικό Τιμόρ 2,5 ε, φορές πάνω, από την ε, ε Ινδία 2,2 δις είναι σήμερα και το 2018 λέει η Παγκόσμια Τράπεζα πρόκειται να ανέλθει σε 4,4 δις δολάρια. Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει συντάξει μια έκθεση ειδική για τη χώρα όπου εκτίθεται ότι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να μην δημιουργηθούν νέοι πόροι, αλλά θα αρκεί η ορθή διαχείριση των υπαρχόντων πόρων. Επίση, λέει η Τράπεζα, πω η ανάπτυξη τη χώρα και τη δυτική Παππού θα πρέπει να γίνει από του κατοίκου τη χώρα. Βεβαίω τώρα υπάρχουν ε, θέματα απόδοση ευθυνών και είπε η Παγκόσμια Τράπεζα ότι τέσσερις από τους 21 δήμους μόνο ε, έκαναν τους οικονομικούς ελέγχους και υπήρξαν ε, συστάσεις όσον αφορά τη χρήση των υπαρχόντων των πόρων, όσον αφορά το σχεδιασμό, προγραμματισμό, <clears throat> τη διαφάνεια, παρακολούθηση κλπ. Επομένως, η τοπική κυβέρνηση ανέλαβε τις ευθύνες ούτως ώστε να εφαρμόσει αυτές τις προτάσεις της διαφάνειας ακριβώς όπως ε, προελέχθη η κεντρική κυβέρνηση. Γι' αυτό το λόγο με μέτρα επετάχυνε την ανάπτυξη της χώρας και υπάρχει το 2007 ένα σφαιρικό ε, πρόγραμμα ανάπτυξης και ε, γι' αυτό και το 2011 επίσης εκδώσαμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές υπάρχει επομένως κάποια ειδική υπηρεσία η οποία συγκροτήθηκε η οποία ε, διευθύνεται από τον κύριο Δελμόνο που κάποτε ήταν ο εκπρόσωπος Ινδονησία στην Επιτροπή Παρακολούθηση Ατσέχ. Και επίση υπάρχει κάποια άλλη ειδική υπηρεσία με τον δόκτωρα Φαρίτ Χουσέιν που είναι ο διαπραγματεύτη μα ε, για τα θέματα ΑΤΣΕΧ. Αν αμφίβολα επομένω έτσι βλέπετε πόσο η κυβέρνηση τη Ινδονησία προτιμά έμπρακτα την επίλυση προγράμματος του προβλήματος, συγγνώμη, μέσω του διαλόγου και ειρηνικά. Τώρα, ο, η ΕΡΕΦΣ Τεμπέη έγραψε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, άρθρο στην τοπική εφημερίδα και λέει ότι πρέπει να δοθεί μια ευκαιρία στην ειρήνη και ότι υπό την αιγίδα του Προέδρου της χώρας έχουν δοθεί νέες ε, δυνατότητες για συνομιλίες ώστε να επιληθεί το πρόβλημα με ειρηνικά μέσα. Πρόεδρε, γενικά η διεθνή κοινότητα και ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να βοηθήσουν. Υπάρχει συμφωνία πλαίσιο και με αυτή τη συμφωνία βέβαια έχουμε διάλογο ανθρώπινα δικαιώματα και υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία μπορούν ε, από κενό να διευθετηθούν και επομένως να συνεχιστούν οι προσπάθειες της κυβέρνησης. Υπάρχει τώρα ένα θέμα μειοψηφία, πλειοψηφία είναι το τελευταίο μου θέμα. Διότι ισχύει το ότι η πλειοψηφία στην Ινδονησία είναι οι μουσουλμάνοι. Όμως είναι μειονότητα μουσουλμάνοι στι ορισμένε περιοχές της χώρας. Διότι έχουμε μία χώρα που είναι α πούμε 80% μουσουλμάνοι, 20% μη μουσουλμάνοι. Στον Παλί 95% είναι Ινδουιστέ, 3% οι μουσουλμάνοι. Στη Βόρεια Σουμάτρα σχεδόν 80% είναι οι χριστιανοί. Στην Παππούα 20% μόνο είναι οι μουσουλμάνοι, 80% είναι οι μη μουσουλμάνοι. Άρα σε μερικά σημεία της ε, χώρας υπάρχει ένα ανακάτεμα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Επομένως, ε, τα, τα πράγματα είναι κάπως πιο περίπλοκα από ότι απλή παράθεση αριθμών. Και ε, όπως προελέχθη σωστά, έχουμε συνεργαστεί δεδομένα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Πολωνική Προεδρία, και εδώ και κάποιες εβδομάδες έχουμε αρχίσει α, τις συνομιλίες για αυτό το πρόβλημα. Πάντως, το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση της χώρας κατανοεί το τι οφείλει να κάνει. Αναγνωρίζει τις ελλείψεις του παρελθόντος και πασχίζουμε για το πώς θα είναι τα πράγματα για όλους καλύτερα στη χώρα και θεωρούμε ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω τώρα που έχει ξεκινήσει ο διάλογος. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πρέσβη, θέλω τώρα να δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας. Δύο λεπτά ο καθένας παρακαλώ, προκειμένου να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα και να κλείσουμε. Παρακαλώ, κύριε Σπάρμπερ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Σύντομα να απαντήσω σε κάποια σημεία που ακούσαμε. Πρώτα απ' όλα για την ειδική αυτονομία. Νομίζω ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους η ειδική αυτονομία απέτυχε είναι ότι δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της Παπούα που είναι περισσότερο πολιτικό παρά οικονομικό. Ο νόμος αυτός για την ειδική αυτονομία που επιτρέπει να δημιουργηθεί η συνέλευση των κατοίκων της Παπούα και την Επιτροπή Συμφιλίωσης κτλ. Η συνέλευση αυτή εξακολουθεί να υπονομεύεται και να είναι αποτυχής. Ό,τι έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ό,τι έχει πάει στα δικαστήρια κλπ. είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν προχωρήσει ικανοποιητικά. Γι' αυτό νομίζω ότι χρειάζονται νέες πρωτοβουλίες που να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των ε, Παππούα, αλλά να το αντιμετωπίζουν ως πολιτικό και να κοιτάνε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουμε περιγράψει. Όσο και το θέμα της μετανάτευσης ε, ή της περιθεροποίησης του πληθυσμού. Για να απαντήσω στην κυρία Γέγκλερ όσον ε, αφορά την κατάσταση ότι δεν είναι δηλαδή σαφής όπως είπε. Και για να απαντήσω επίσης και στο σχόλιο του Προέδρου για τη δυσκολία πρόσβασης, αυτό είναι στοιχείο κλειδί. Και άρα λοιπόν η ιδέα του να πάει μία αντιπροσωπεία της υποπιτροπής αυτής ή κάποιες άλλες επιτροπής στη Δυτική Παπούα για λόγους ερευνητικούς θα ήταν κάτι που θα βοηθούσε πράγματι πολύ. Και αυτό θα ήθελα να καταγραφεί παρακαλώ. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, η Δόκτωρ Κόρπεκ. Αγαπητέ πρέσβη, θέλω να πω ότι συμφωνώ και παραυξάνω τόσα υποπρολαλή σας, ότι δηλαδή δεν είναι δυνατόν να λυθεί το πρόβλημα με τον νόμο αυτό, ο οποίος έξι χρόνια υπάρχει αλλά δεν φέρνει αποτελέσματα. Τον υπόσχεστε δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Ο ειδικό νόμος αυτονομίας τελικά ήδη από το 2001 μέχρι το 2006 δεν βοήθησε τους κατοίκους να προσφέρουν αυτή κάτι. Και αυτό γιατί, γιατί η εντολή είναι τέτοια όσον αφορά την Επιτροπή Συμφιλίωσης στην Παπούα και στην Άτσε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν φέρνει αποτελέσματα. Αυτό που μπορεί να γίνει στην Παπούα και στην Άτσε είναι μόνο οι οικονομικές ε, δεχομένως από ζημιώσεις, τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν θέλω να κάνω έκκληση προς την κυβέρνηση της Ινδονησίας να εφαρμόσει κάτι το οποίο έξι χρόνια έχει υποσχεθεί τώρα. Δεύτερον, όλοι εδώ συμφωνήσαμε, από ό,τι έχω καταλάβει, για το ότι ο διάλογος είναι κάτι που θέλουμε. Και επιτέλους ο πρόεδρός σας μίλησε για διάλογο. Ε, του πήρε χρόνο. Πέρασαν διάφορες θητείες, έγιναν διάφορες ανακοινώσεις. Όντως, εκτιμούμε όλους ιδιαίτερο τη λέξη διάλογο που πρόφερε. Όμως οι διάφοροι οι οποίοι ορίζονται για την μονάδα αυτή δρούν με διαφορετικούς τρόπους. Ο Πάντανα μόνο πηγαίνει προς μία κατεύθυνση, ο Δόκτωρ Βάρικο πάει προς μια άλλη κατεύθυνση. Οπότε έχουμε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις οι οποίες μάλλον ανάποδα αποτελέσματα φέρνουν. Και γι' αυτό δεν έχει υπάρξει καμία πρόοδος η ομάδα αυτή δεν έχει καν φτιαχτεί. Φανταστείτε πόσο δύσκολο θα είναι να λειτουργήσει κιόλα. Ευχαριστούμε κύριε Κόρβερ. Λέω πρόεδρος, κυρίες και κύριοι. Παρατείναμε για ένα τέταρτο το χρόνο που είχαμε προβλέψει να αφιερώσουμε στο θέμα της Παπούα και της Δυτικής Παπούα. Σίγουρα κατά τη διάρκεια αυτή τη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα επανέλθουμε ξανά και ξανά. Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι εύκολο να λυθούν τα προβλήματα τα οποία έχουν τις ρίζες τους βαθιά στο παρελθόν. Προβλήματα τα οποία δεν λύθηκαν στα μάτια του τοπικού πληθυσμού. Πάντως πρέπει να αναλάβουμε ό,τι δράση μπορούμε για να πετύχουμε το στόχο μας. Θέλω εδώ να πω ότι οι εκπρόσωποι της αντιπροσωπείας ΑΣΕΑΝ δεν μπόρεσαν να έρθουν σήμερα εδώ. Η γραμματεία όμως, η γραμματεία τους είναι εδώ και η γραμματεία τους θα φροντίσει και θα συμμετάσχει στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Βερμπέρ και την ε, κυρία Κόρβερ και τον Τώρα περνάμε στην ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την Βιρμανία. Την τελευταία φορά, το Μάιο, μιλήσαμε για αυτό το θέμα και από τότε είχαμε μεγάλες αλλαγές στη χώρα, τις οποίες θα πρέπει και να συζητήσουμε. Γι' αυτό ακριβώς αποφασίσαμε να έχουμε στην ημερήσια διάταξη αυτό το θέμα. η κυρία Αουν Σαν Σουκή, από ό,τι φαίνεται, θα είναι υποψήφια στις ε, νέες εκλογές. Θα θυμόσαστε, δίχως άλλο, ότι η προηγούμενη νίκη του κόμματός στις εκλογές δεν αναγνωρίστηκε από, την, ε, από το στρατιωτικό καθεστώς εκεί. Όμως, οι αρχές προχώρησαν σε μεταρρυθμίσεις με τις οποίες είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη η διεθνής κοινότητα. Η Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, η ίδια η κυρία τον πήγε στην ε, Βυρμανία και η δική μας ΑΣΕΑΝ αποφάσισε επίσης να έχει μια αντιπροσωπεία εκεί. Η κυρία Άστον, από τη δικιά της την πλευρά, δηλώνει πολύ ικανοποιημένη από το γεγονός ότι οι αρχές έδωσαν αμνηστία σε ένα μεγάλο μέρος των πολιτικών ε, κρατουμένων. Εννοείται ότι θέλουμε να απελευθερωθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι. Θέλω λοιπόν να έχουμε καταρχήν το βίντεο, να το δούμε, για να μπορέσουμε και να ακούσουμε έτσι την δήλωση της κυρίας Aung San Είναι μια δήλωση που έκανε ε, την στιγμή που είχαμε την τελετή για την απονομή του βραβείου Σαχάροφ. Μας μιλάει λοιπόν και για τη σημασία που έχει το βραβείο Σαχάροφ και που είχε και στο παρελθόν για το μέλλον της ε, Γερμανίας. Σας είμαι ε, ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνετε να μεταφέρω το μήνυμα μου αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή που είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι στην καρδιά όλων ημών που δουλεύουμε για τη δημοκρατία στη Βερμανία. Ακριβώς επειδή παραβιάζονταν τα ανθρώπινα δικαιώματα, γι' αυτό και εμείς αγωνιζόμαστε τόσο καιρό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας έχει βοηθήσει στον αγώνα μας αυτό. Η δικιά σας στήριξη και η δικιά σας κατανόηση είναι αυτά τα οποία μας έφεραν φως μέσα στις σκοτεινές μέρες όπου ήμασταν αντιμέτωποι με τόσο σκληρή καταπίεση, τόσο που νομίζαμε ότι δεν θα μπορούσαμε να τα βγάλουμε πέρα ποτέ. Όμως η ελπίδα μας δεν μειώθηκε ποτέ γιατί ξέραμε ότι είχαμε φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, φίλους και συμμάχους οι οποίοι ήταν έτοιμοι να μας στηρίξουν. Και είναι μια σημαντική σύμπτωση το γεγονός ότι το βραβείο Ζαχάροφ απενεμήθη σε μένα σε μια στιγμή όπου εμείς το κίνημα για τη δημοκρατία στην ε, Βυρμανία αντιμετωπίζαμε πραγματικά μεγάλες δυσκολίες. Ήταν η στιγμή που μας ε, φαινόταν ότι ο κόσμος μας είχε ξεχάσει. Ήταν η στιγμή όπου νομίζαμε ότι ήμασταν μόνοι μας στον ε, αγώνα. Αλλά το βραβείο Ζαχάροφ, το οποίο απενεμήθη σε μένα, απενεμήθη σε μένα όχι σαν άτομο, αλλά σε όλους εμάς που αγωνιζόμαστε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βυρμανία. Και μας θύμισε ότι δεν είμαστε μόνοι. Ξανά ε, και ξανά το θυμόμαστε αυτό. Θυμόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι, ότι δεν μας έχετε ξεχάσει. Για άλλη μια φορά λοιπόν θέλω να σας πω ότι είμαι ευγνώμων σε ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλα όσα έκανε αυτό προκειμένου να κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες μας και να σας πω επίσης ότι περιμένουμε ανυπομονησία την ημέρα εκείνη που θα μπορέσουμε να βρεθούμε πιο κοντά ως φίλοι και ως σύμμαχοι, δουλεύοντας μαζί για έναν περισσότερο ασφαλή και ευτυχισμένο κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ όντως το βραβείο Ζαχάροφ αυτό γιατί για πολλά χρόνια κατά τη διάρκεια δηλαδή τόσων διώξεων δεν έχασε ποτέ την ελπίδα της και περιμένει με ανυπομονησία όπως λέει την μέρα εκείνη που θα μπορέσει πραγματικά να αναλάβει δράσεις για να αλλάξει η κατάσταση στη Βυρμανία. Ελπίζουμε ότι η μέρα αυτή θα έρθει. Όλα αυτά δείχνουν πόσο επηρεάζει τελικά τα πράγματα το βραβείο Ζαχάροφ που αποτελεί μια μεγάλη ηθική στήριξη για όλους όσους υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μας ε, έδειξε και πόσο μετριόφρον είναι όταν είπε ότι το βραβείο αυτό δεν απενεμήθη μόνο σε εκείνην προσωπικά, αλλά σε όλους όσους αγωνίζονται και είναι ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα αυτή. Θέλω τώρα να ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Ο κύριος Γκίλεσπη. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όντω οι τελευταίοι μήνε στη Γερμανία ήταν σημαντικοί. Τον Νοέμβριο που μας πέρασε, όταν έγιναν οι εκλογές εκεί, δεν ήταν ελεύθερε οι δίκαιε εκλογές, δεν μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε έτσι. Όμως, σιγά σιγά όλοι το κατάλαβαν, υπήρξε απογοήτευση. Μέσα στου επόμενου όμως μήνε άλλαξαν τα πράγματα σημαντικά. θα έλεγα μετά την ομιλία του Προέδρου που έκανε τον Απρίλιο στο Κοινοβούλιο, όπου εκεί έθεσε μια σημαντική μερίσια διάταξη και δεσμεύτηκε να την τηρήσει με διάφορα σημεία μεταρρυθμίσεων, στα οποία περιλαμβάνονται και πράγματα όπως είναι προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταπολέμηση της διαφθοράς και αντιπολίτευση και εθνοτικές ομάδες. Τότε είπαμε ότι ίσως τα είπε αυτά έτσι για να τα έχει πει. Αλλά αναλύοντας τη γλώσσα και τα διάφορα σημεία καταλάβαμε ότι τενούσε. Και έκτοτε είχαμε νέες εξελίξεις πράγματι που όλες πηγαίνουν προς την ίδια θετική κατεύθυνση. Εννοείται ότι έχουμε κοιτάξει πάρα πολύ την περίπτωση της αντιπολίτευσης, τις επαφές με την κυβέρνηση, την ε, τροποποίηση επίσης για την καταγραφή των πολιτικών κομμάτων και του NLD, της Aung San Suu Kyi, που νωρίτερα δεν ήθελαν να τον αναγνωρίσουν. Τώρα όμως αποφάσισε το κόμμα αυτό να συμμετάσχει στις εκλογές που θα λάβουν χώρα του χρόνου και όπου θα συμμετέχουν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πίσω όμως από αυτές τις εξελίξεις που είναι έτσι τόσο εμφανείς, έχουν υπάρξει και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα ε, που έχουν γίνει στο Κοινοβούλιο με σχέδια νόμου και ένα από τα πρώτα που πέρασε ήταν ένας νόμος που επιτρέπει τα συνδικάτα. Νομοθεσία η οποία επίσης απαγορεύει ε, την δουλεία, θα περάσει σύντομα από το Κοινοβούλιο και άλλα. Συγχρόνως ο πρόεδρος επανέλαβε την επιθυμία του να συζητήσει επικοδομητικά με διάφορες εθνοτικές ομάδες για να καταλήξουν σε ειρηνικές συμφωνίες. Μέχρι τώρα έχει υπάρξει κάποια επιτυχία στο κρατήριο σαν παράδειγμα, αλλά η πρόκληση εξακολουθεί να παραμένει. Υπάρχουν συγκρούσεις σε διάφορες περιοχές αλλά αν μη τι άλλο, οικονομικά και πολιτικά θα λέγαμε ότι αντιμετωπίσει καλύτερα τα αιτήματα των εθνωτικών ομάδων η κυβέρνηση από ό,τι κατά το παρελθόν. Όλα αυτά λοιπόν είναι θετικά. Τώρα, τι πιστεύουμε. Είναι, ξεπερνάει τις προσδοκίες μας. Όλοι είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Όλοι βέβαια ρωτιόμαστε για την ποιότητα των αλλαγών και πόσο θα κρατήσουν οι αλλαγές αυτές. Και όταν μιλάω για την ε, ποιότητα των αλλαγών, ε, προς Θεού δεν θέλω να μειώσω τη σημασία των γεγονότων, απλώς αναρωτιέμαι κάποια πράγματα. Κοιτάμε την ομοθεσία, λοιπόν. Γενικά, τα νομοσχέδια που προτείνονται είναι καλά. Αυτό για τα συνδικάτα όντως ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές ε, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Τώρα άλλε μεταρρυθμίσει που προτείνονται επικεντρώνονται κυρίως στην αγροτική μεταρρύθμιση και σε ειδικά θέματα που έχουν να κάνουν με την, με την μικροχρηματοδότηση των αγροτών. Θα μπορούσαν να υπήρχαν περισσότερα πράγματα για την κατανομή της γης, αλλά φαντάζομαι ότι θα γίνει και αυτό εν καιρό. Τονίζεται λιγότερο ίσως ο τομέας των επιχειρήσεων και των επενδύσεων. Είναι κατανοητό αλλά θα θέλαμε να ξεκινήσει και αυτό μέσα στην επόμενη περίοδο. Επίσης, για τις αλλαγές. Αυτό το νέο σύστημα με το Σύνταγμα του 2008, το σύστημα δηλαδή των περιφερειακών κοινοβουλίων, κυβέρνηση, στρατού κτλ. Όλα αυτά ξεκινάνε από τη στρατιωτική κυβέρνηση βέβαια, οπότε η καλύτερη ερμηνεία μας ήταν ότι έγιναν για να ε, μπορέσει να υπάρξει έλεγχος ε, στις αλλαγές από την απερχόμενη στρατιωτική κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνουν κάποια όρια στις μεταρρυθμίσεις βραχυπρόθεσμα. Και στη συνέχεια έχουμε να κάνουμε και με εντάσεις που υπάρχουν μέσα στην κυβέρνηση για το βηματισμό, για το ρυθμό και την έκταση των μεταρρυθμίσεων. Δεν πρέπει βέβαια να σκεφτούμε ότι από τη μια έχουμε του μεταρρυθμιστέ και από την άλλη μεριά έχουμε του σκληροπυρηνικού. Όχι. Πρέπει να σκεφτούμε τι είναι αυτό που πιέζει για μεταρρυθμίσεις, ποιος θα υποφεληθεί από αυτές και ποιος αντίθετα υποφελείται από το παλιό σύστημα. Άρα στην κυβέρνηση υπάρχει κάποια ένταση. Και εμείς λέμε ότι αυτή η ένταση οδηγεί σε κάποιο περιορισμό ε, του ρυθμού με τον οποίο προχωράνε οι μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να είμαστε βέβαια ρεαλιστέ για το ότι είναι εφικτό. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι λογικό να περιμένουμε κάποια πράγματα να συμβούν τα οποία θα υπονομεύσουν την σοβαρότητα με την οποία προχωράνε οι μεταρρυθμίσεις. Τι θα ήταν αυτό είναι το θέμα του αριθμού των πολιτικών ε, κρατουμένων. Το κόμμα NLD μίλησε για 700 αλλά πιστεύουμε ότι το νούμερο είναι μεγαλύτερο. Μέχρι 2.000. Τώρα μπορεί το 2.000 να είναι μεγάλο νούμερο, αλλά ίσως είναι 1.000, 1.200. με πολιτικούς κρατουμένους από εθνοτικέ ομάδε. Τώρα 200 απελευθερώθηκαν, οπότε περιμένουμε εμεί κάτι πιο ουσιώδες να γίνει. Ελπίζουμε. Έπειτα οι εκλογέ ελπίζουμε ότι θα είναι πιο ελεύθερες, πιο δίκαιες από ό,τι ήταν εκείνες που είχαμε το 2010, τον 2010. Ο πρόεδρος είπε ότι αυτό είναι ο στόχος του. Ελπίζουμε να το δούμε και η αντιπολίτευση και το κόμμα NLD να έχουν όλες τις ευκαιρίες που μπορούν για να προχωρήσουν. Μέσα στο επόμενο εξάμεινο, πιστεύω, θα δούμε το διάλογο ανάμεσα στην κυβέρνηση και την ούσα Σουική να λαμβάνει χώρα. Όπως επίσης και με τα άλλα ε, πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Ξέρουμε ότι υπάρχουν καλές επαφές ανάμεσα σε πολιτικούς από το κυβερνών κόμμα και την αντιπολίτευση και ελπίζουμε αυτό να αποκτήσει πιο βαθιές ρίζες και να διαρθρωθεί σιγά σιγά αυτός ο πολιτικός διάλογος για το μέλλον της χώρας. Αλλά επαναλαμβάνω κατόπιν τούτων ότι με τίποτα δεν θέλω να μειώσω τη σημασία που έχουν τόσα έγιναν μέχρι τώρα. Όμως θα ήθελα να δούμε και αυτή τη συνέχεια για να μπορέσουμε να πούμε ότι η πολιτική αλλαγή στη Βερμανία είναι κάτι ουσιαστικό, είναι κάτι το οποίο, στο οποίο μπορούμε να ανταποκριθούμε και εμείς θετικά. Εμείς από την πλευρά μας συνεχίζουμε την διαδικασία που έχουμε αναλάβει ανάλυσης των ε, γεγονότων για ένα μήνα ακόμα θα το κάνουμε και από εκεί και πέρα ε, θα δούμε με το Συμβούλιο βέβαια που συνήθως βάζει περιορισμούς ε, θα δούμε και εμείς από την πλευρά μας βάσει των θετικών αλλαγών που θα δούμε ακόμα πώς θα αντιδράσουμε. Συγχρόνως όμως κάτι το οποίο μας απασχολεί πολύ είναι το θέμα της εφαρμογής των όσων κάνει η κυβέρνηση, δηλαδή φτιάχνοντας αυτό το σώμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πόσο αποτελεσματικό θα είναι θα εξαρτηθεί από τις δυνατότητες που θα έχει να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις και ξέρουμε ότι υπάρχουν αδυναμίες στο σύστημα. Προκειμένου και να καθοριστεί σωστή πολιτική και να τεθεί σε εφαρμογή. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά τον καθορισμό ορμοδιοτήτων των περιφερειακών κοινοβουλίων και τις σχέσεις τους με την κεντρική κυβέρνηση. Άρα, η οικοδόμηση ικανοτήτων είναι κάτι που μας απασχολεί όλος ιδιαίτερος και πιστεύουμε ότι επήγει όπως επίσης και η αύξηση των πολιτικών επαφών, ώστε να στείλουμε το μήνυμα που να λέει ότι εκτιμούμε όλους ιδιαίτερως τα όσα συμβαίνουν και περιμένουμε να πάνε ακόμα πιο μακριά. Ώστε μήπως και το σε μπορέσει να δραστηριοποιηθεί, δίνοντας τεχνική αρρωγή για τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις με συμμετοχή και του Διεθνούς Μεσολατικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζης. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι είμαστε πολύ θετικοί, περιμένουμε να προχωρήσουν ακόμα περισσότερο, ώστε να φανεί ότι είναι μια πραγματικότητα και από εκεί και πέρα θα φροντίσουμε και εμείς να τα αποκριθούμε με τον κατάλληλο τρόπο. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γκυλέσπη. Να δώσουμε τώρα την επικεφαλής του Γραφείου για τη Βερμανία της Ευρώπης, την ε, κυρία Κόλεν. Ευχαριστώ. Ο ακλαστικός διευθυντής μας ε, θα ήθελε πολύ να είναι παρόν σήμερα. Βεβαίως ε, δεν μπορούσε σήμερα να είναι εδώ, οπότε θα διαβάσω εγώ το μήνυμα, το μήνυμά του. Παρά το ότι παρατηρώ ότι με το μεγαλύτερο μέρο τη επαγγελματική ζωή μου την κατάσταση στην Βερμανία, πρώτη φορά ε, γύρισα, επέστρεψα από το πρώτο μου ταξίδι ε, εδώ και 50 χρόνια στη Βερμανία. Ε, από το 1962, εγώ που ήμουν μικρό, τότε ξεκίνησε η κατάληψη της Βερμανία και τότε είχε ανακοινωθεί ότι όντω ε, θα μπορούσαν οι πρόσφυγες να ε, επιστρέψουν και ήθελα να δω κι εγώ τι έγινε και να δω την, ε, το σπίτι μου. προσπάθησα να συναντηθώ και τα κατάφερα με εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, με, τη, με κυβερνητικούς αξιωματούχους. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου είδα ότι η πολιτική ατμόσφαιρα είναι πολύ αισιόδοξη και πιο ανοιχτή από ό,τι περίμενα οι πολιτικοί, οι πολίτες ε, φαίνεται ότι φοβούνται λιγότερο πια. Υπήρχε μεγάλο σκεπτικισμός για τις εκλογές και τη νέα κυβέρνηση μέχρι το τέλος του Ιουλίου του τρέχοντος. Και εγώ ήμουν πολύ σκεπτικός και εξεπλάγινα από την ε, ε, ομιλία του Πρωθυπουργού που ανακοίνωσε μία μεταρρυθμιστική ατζέντα. Ε, και ξαφνικά τον ε, Αύγουστο όλα ε, ξεκίνησαν να κινούνται προς τα, μπρο, προς τα μπρος. Ο Πρωθυπουργό συναντήθηκε με την Αούγκ Σανσουκή, η οποία ήταν θετική και είπε ότι θα πρέπει οι εξόριστοι να επιστρέψουν. Άρχισαν να γίνονται συζητήσεις με εθνοτικές ομάδες. Ο πρόεδρος ξεκίνησε διαδικασίες κοινοβουλευτικών συζητήσεων οι οποίες δημοσιεύονται και το εύρος της συζήτηση ήταν ιδιαίτερα μεγάλο, με, ακόμη και για ευαίσθητα θέματα όπως εθνική συμφιλίωση, αμνηστία, απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, πυρηνικά προγράμματα, θέματα δηλαδή που θα ήταν τελείως αδύνατο να συζητηθούν υπό τα προηγούμενα καθεστώτα. Δημιουργήθηκε μια Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επίσης νέα εργατική νομοθεσία για το συνδικαλισμό. Κάποιοι πολιτικοί κρατούμενοι επίσης απελευθερώθηκαν. Η κυβέρνηση αναθεώρησε τον ε, εκλογικό της νόμο για να μπορέσει να καταγραφεί, να καταχωρηθεί και το NLD και το NLD τώρα έχει ε, καταχωρηθεί ως πολιτικό κόμμα και θα συμμετάσχει στο το 2015 στις εκλογές. Η Aung San Suu Kyi έχει προτείνει ότι μπορεί, έχει προτεθεί να είναι υποψήφια για τις ε, εκλογές που θα γίνουν τον επόμενο χρόνο. Δεν μπορώ να μιλήσω για το μέσο πολίτη, αλλά αισθάνομαι ότι οι άνθρωποι που συνάντησα έχουν όντω την εντύπωση πω τα πράγματα έχουν αλλάξει. Σε ό,τι αφορά τι εθνικέ διαμάχε, οι περισσότεροι, ε, και η διεθνή κοινότητα, θεωρούν ότι το πρόβλημα αυτό είναι περιφερειακό. Θεωρούν ότι μόλι έχουμε, την δημοκρα... έχουμε εγκατάσταση δημοκρατία, το πρόβλημα αυτό θα λυθεί στη Βυρμανία. Αυτό όμω δεν είναι αληθέ το πρόβλημα προκύπτει από τον καιρό της δημοκρατίας στη χώρα. Η Βρυμανία έχασε τη δημοκρατία της και την ελευθερία της γιατί δεν υπήρξε συμφωνία για το πώς προσπαθούσε η δημοκρατικώς εκλεγμένη κυβέρνηση να ε, συντάξει, να εφαρμόσει την πολιτική της αλλάζοντας το Σύνταγμα. Ένας πιθανός δρόμος για να προχωρήσουμε θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε τις ε, προβλέψεις του συντάγματος ε, του 2008 που επιτρέπει ε, κρατικές, τις κρατικές κυβερνήσεις. Η εντολή αυτή είναι περιορισμένη βεβαίως αυτών των σχηματισμών, αλλά είναι το μόνο σύνταγμα που υπάρχει και το οποίο ασχολείται με το θέμα αυτό της αυτοδιάθεσης την οποία ζητούν τα, οι διάφορες ε, από, ε, από τον καιρό τη ανεξαρτησία. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα, μια παράλληλη διαδικασία με την διαδικασία αποκέντρωσης. Ε, εγώ συνάντησα πολλούς και οι οποίοι ήταν πολύ προβληματισμένοι για την δυνατότητα της κυβέρνησης να λειτουργήσει. Γιατί η μηχανή ακόμη λειτουργεί με τους παλιούς κανόνες, ενώ πολλοί θέλουν να υπάρξει αλλαγή. Ποια, τι θα μπορούσε λοιπόν η διεθνή κοινότητα και εσεί ω κοινοβουλευτικοί να κάνει. Θα μπορούσατε να δώσετε την υποστήριξή σα για τη βελτίωση αυτών των δημοκρατικών θεσμών που υπάρχουν. Ο πρόεδρο λέει ότι είναι υπόλογο στο Σύνταγμα. Θα πρέπει να τον ενθαρρύνουμε ώστε να. Ε, συντάξει, να, εξασκεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με το ε, Σύνταγμα. Να, κάνει την, να όντως να δημιουργήσει ένα κράτος δικαίου αντί να ε, διοικεί με, τον, ε, με τους αυθαίρετους κανόνες ενός δικτάτορα. Θα πρέπει να, οι υποψήφοι και οι βουλευτές που θα εκλεγούν να είναι υπόλογοι στον λαό που τους εξέλεξε. Αν θέλουμε μια βιώσιμη δημοκρατία, τα πολιτικά κόμματα πρέπει να είναι δημοκρατικά και στην δομή και στις πολιτικές τους. Πρέπει να τους βοηθήσουμε να βελτιώσουν τη δυνατότητα για εκπόνηση πολιτικής, για χάραξη νομοθεσίας και για την παρουσία του οράματός τους στον, στο ευρύ κοινό. Οι δημόσιοι υπαλλήλοι επίσης πρέπει να εκπαιδευτούν για να είναι πιο αποτελεσματικοί στην ε, εκτέλεση των καθηκόντων τους αντί να υποκύπτουν κάθε φορά στις ε, επιθυμίες ενός ε, αυτοκρατορικού ηγέτη εισαγωγικά. Ε, πρέπει λοιπόν το σύστημα να γίνει δημοκρατικό και για να γίνει αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε ε, πιθανότητα υπάρχει για να προωθήσουμε δημοκρατικά ιδεώδη και πρακτικέ στα πλαίσια της κυβέρνησης έτσι ώστε να μπορέσουν να θεσμοθετηθούν και να μην ε, μπορούν να ανακληθούν. Αν θέλουμε η Βερμανία να αποτελέσει ένα ιδεατό δημοκρατικό κράτος, προφανώς πολύ απέχουμε ακόμη ε, από αυτό και βεβαίως ε, θα εξαρτηθεί το πόσο γρήγορα θα φτάσουμε σε αυτό το όραμα. Αλλά αν μπορέσουμε να συγκρίνουμε το τι γίνεται τώρα στη Βερμανία με το τι γινόταν πριν από 6 μήνες, σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι τα πράγματα όντω αλλάζουν. Ευχαριστώ. Dziękuję pani a jednocześnie dziękuję również panu Harnie ο Πρόεδρος. Και εγώ με τη σειρά μου τον ευχαριστήσω τον uh, κύριο Γιάνκοβε, ο οποίο δεν μπόρεσε να παραστήσει στη συνάντησή μας, αλλά μας διεβίβασε το μήνυμά του. Όχι, εδώ και πολύ καιρό. Δεν έχουμε ακούσει τέτοια, τόσα θετικά εδώ στην Επιτροπή μας. Informacje o tych zmianach i sądzę, że to jest bardzo dobra e, informacja ze strony państwa, ale jednocześnie też i troska czy ten proces jest procesem trwałym. Επομένω, έχουμε αυτή την ενημέρωση για τόσα γίνονται στι χώρε ε, αυτών των αγωνιστών και ε, βεβαίω το θεμητό είναι να δούμε κατά πόσον οι αλλαγέ οι οποίε αχνοφέρονται κατά πόσον θα παγιωθούν. Και τώρα να καλέσουμε με τη σειρά του τον ε, κύριο πρέσβη, εάν θέλει να λάβει τον λόγο. Ε, Α, δεν είναι εδώ takiego, takiej chęci, więc chciałem zapytać pana ambasadora Timansa oraz pana... Όχι, δεν θέλει το λόγο. Κύριε Γκυλέσπε, κύριε Τίμενς, ποιος θέλει να λάβει το λόγο. My experience of dealing with, um... Η δική μου εμπειρία από την αναμέτρηση με τη γραφειοκρατία. Όχι, δεν οδηγεί σε αδιαφορία ούτε σε αδράνεια γιατί έχουμε αυτούς τους τρεις εξαίρετους διπλωμάτες. Ένας εξ αυτών τώρα έγινε υπουργό εξωτερικών και εδώ και κάποια χρόνια αρχίσαμε διστακτικά τον διάλογο με την κυβέρνηση της χώρας όσον αφορά την καταπολέμηση της παινίας σε τρεις ε, τομείς για στέγαση, συνθήκες διαβίωσης, γενική πρόνοια και υπήρχε συμμετοχή από Αυστραλία, από Ευρώπη, από Αμερική, από πανεπιστημιακούς ε, και παρά τις δύσκολες συνθήκες ε, υπήρχε μεγάλη προθυμία οπότε θεωρώ ότι πάντα δυσκολίες ε, αφού μπορούμε να καταφέρουμε αυτή την προσπάθεια, η κυβέρνηση και η διοίκηση μπορούν να σημειώσουν πρόοδο όσον αφορά την ανάπτυξη της χώρας. Και με τις μεταρρυθμίσεις θα αποδείξουν ότι μπορούν να κάνουν τη διαφορά όσον αφορά την ευημερία του λαού. Και εμεί βαθιά προβληματιζόμαστε για το τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τα πράγματα. Πάντω, εάν η διεθνή κοινότητα μπορεί να εμπλακεί περισσότερο, θα είναι θετικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο άλλος διπλωμάτης κύριος. Και εγώ ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να πω σε συνέχεια τον όσον είπε ο συνάδελφος ε, ο Σέμος ότι είναι κάποιο που ξέρει βαθιά τα θέματα της χώρας. Εγώ, αντίθετα με εκείνον, δεν έχω πατήσει ποτέ μου εκεί. Δεν παρουσιάστηκε ευκαιρία. Είναι γνωστέ δυσκολίε όταν υπάρχουν τέτοια κατεπιστικά αυταρχικά καθεστώτα και σε συνέχεια των όσων υποσέμουν και και εμεί θεωρούμε ότι είναι εξελίξει πάρα πολύ θετικέ και ότι. Έτσι. Έχουμε ξεκινήσει την ομάδα επαφών για τα θέματα των δικαιωμάτων. Ακόμα βέβαια δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδο. όμως νομίζω ότι τώρα προσπαθούμε να δούμε τι εναλλακτικέ υπάρχουν τόσο ώστε να μπορέσουμε τις ε, μεταρρυθμίσεις να τις υποστηρίξουμε και επίσης θα οργανώσουμε και κάποιες ε, αποστολές να δούμε και τι θα αποδώσει και η επίσκεψη της Χίλαρη Κλίντον. Νομίζω, νομίζω θα επηρεάσει τα πράγματα. Και σε επίπεδο η Αστυνία Υόρκη. Κάνουμε κάποια διαβήματα και εκεί πέρασε κάποιο ψήφισμα για τη χώρα. Προσπαθήσαμε να προσαρμοστούμε στις συνθήκες που αλλάξανε. Πάντως τελικά τα συμπεράσματα μοιάζουν με αυτά στα οποία κατέληξε ο ύπατος εκπρόσωπος ότι ακόμα υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Και θα πρέπει να συγχυστούν οι προσπάθειες. Και εμείς θα κατάλαβουμε προσπάθειες από δική μας πλευράς για να βοηθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Επίση. δεν πρέπει να έχουμε ψευδεστήσει. Ξέρουμε τι έχει γίνει στην περιοχή αυτή. Πάρα πολύ δύσκολη η πρόοδο και το να αποσπάσει κανεί ε, στέρε δεσμεύσει, ιδίω όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και να, αποσπάσει κανεί μια, μια ουσιώδη δεν είναι τόσο δύσκολο. Και τελικά να υπάρξει ουσιαστικό διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ινδονησία, Βιετνάμ, Καμπότζη. Πάντω τον Ιανουάριο θα αρχίσει με τέτοια προσπάθεια. Πάντω από αυτό μέχρι το να διαπιστώσει κανεί σε κάποιε ουσιαστικέ αλλαγέ, ε, αυτό είναι διαφορετικό. Και πάντοτε εξαρτάται από την θέληση των όσων έχουν τα ενία της εξουσίας. Οπότε γι' αυτό σας λέω ότι θα πρέπει να θεωρηθεί όχι ειδωμένο απομονωμένο των δικαιωμάτων, θα πρέπει να ειδωθεί ή στο πλαίσιο της γενικότερης εξέλιξης ανάπτυξης της χώρας και της υποχρέωσης ε, λογοδοσίας μιας κυβέρνησης. Ο πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Τίμανς. Κυρίες και κύριοι, κατόπιν των όσων ε, ακούσαμε, δεν μπορούμε παρά να θεωρούμε ότι οι θετικές αυτές θα γίνουν μια εξελικτική διαδικασία θετική για τη χώρα. Και θα συνεχιστεί η πρόοδος και ότι θα επηρεαστούν οι αρχές της χώρας από τις θετικές εξελίξεις σε άλλες χώρες, φερειπίνες στη δική μας χώρα, τις οποίες ο ΙΠΕΞ μετέβη στην Γερμανία. Απάντησε σε πολλές ερωτήσεις και θεωρώ ότι το ενδιαφέρον των αρχών στο δημοκρατικό μετασχηματισμό είναι καλά μαντάτα. Άρα αξίζει κανείς να ενημερώνεται για τις δημοκρατικές εξελίξεις σε άλλες χώρες από τη δική του, για την αλλαγή σε πολλές Επίση Επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι οι δηλώσεις Κοέν σημαίνουν ότι υπάρχουν και από, την, και από το μέτωπο της, της μετανάστευσης θετικά Να ευχαριστήσουμε όλους τους καλεσμένους μας, όλους όσοι θέλησαν να μας βοηθήσουν να εξαντλήσουμε τη μέση διάταξη. Ευχαριστούμε για τα συμπεράσματα, ευχαριστούμε την εξωτερική υπηρεσία το Συμβούλιο. Οπότε τώρα θα κάνουμε διάλειμμα στις τις 3 ώρες. Ευχαριστούμε και τους διερμηνείς. Θα τα ξαναπούμε στις 3. Θα συνεχιστεί η συζήτηση. Θα συζητήσουμε με τον κύριο Ποπόφσκι και θα γίνει μια σχετική ενημέρωση.